So, good morning, everybody. I think um, we've rescued Mr. Hatsimakakis from the traffic jam. Καλημέρα σας. Ευτυχώς γλιτώσαμε από την πρωινή κίνηση και είμαστε παρόντες για να ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την πρόσβαση στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ε, εισηγητή Γιώργο Χατζημαρκάκη που ρύθμισε και την παρουσίαση ώστε να ζωντανέψει το νομικό κείμενο, κάτι το οποίο είναι πολύτιμο Συχνά τα νομικά κίνημα είναι πολύ στεγνά και δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε παραδείγματα για το τι ακριβώς εννοούν. Θα ακούσουμε λοιπόν τους προσκεκλημένους σου σε λίγο. Και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Τσαφκόφσκι, τον κύριο Ραμόν, την κυρία Ρούλε. Εγώ είμαι σκιώδης για την ομάδα μας και αλλιώς. Έχουμε λοιπόν εκπροσώπους των διαφόρων ομάδων που θα συμμετέχουν στη συζήτηση. Το λοιπόν, ο Γιώργος Χατζημαρκάκης. Θα, ε, θα συστήσεις εσύ τους προσκεκλημένους. Έχω τα ονόματά τους, αλλά νομίζω πως θα ήθελες εσύ να τους συστήσεις και να κάνεις και την εισήγηση για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε να κάνουμε αυτή την παρουσίαση που ε, θα μας τονώσει τη μνήμη διότι Mm-hmm. Μπορεί να ακούγεται πολύ τεχνικό αυτό το θέμα της νομοθεσίας, αλλά αυτό το νομοθέτημα ε, θα το λέω στα εγγόνια μου ότι ήμουν εισηγητής, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πολλούς. Εγώ θα έλεγα κάποια μέρα για όλους μας. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε δυσκολίες εμείς να μπούμε σε ιστοτόπους. Αργότερα θα μπούμε στην ουσία του θέματος. Το μόνο που θέλω να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή είναι να καλωσορίσω ορισμένους ε, καλεσμένους μας που θα μας ε, πούν αλλά και θα μας δείξουν πόσο δύσκολο είναι να παρακάμψει κανείς αυτό το πρώτο εμπόδιο. Για κάποιον που έχει αναπηρία, για κάποιον που χρειάζεται πληροφορία. Και αυτό το πρώτο εμπόδιο είναι ακριβώς το εμπόδιο ε, να μπει στην πληροφορία. Η πρώτη ψυχρολουσία. Όλα τα άλλα εμπόδια, αν θέλει κανείς, ας πούμε, ε, όταν θέλει να πάρει ένα λεωφορείο, έχεις πολλά προβλήματα, αλλά πρέπει να ξέρεις τι ώρα φεύγει, πού βγάζει εισιτήριο, πώ το πληρώνει. Και αυτό το πρώτο εμπόδιο, το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο που βγαζει εισιτηριο πως το πληρωνεις και αυτο το πρωτο εμποδιο το πρωτο βημα ειναι το σημαντικοτερο που πρεπει να γίνει. Λοιπόν, αυτό συζητούμε τώρα, πώς θα ξεπεραστεί η αρχική δυσκολία. Ε, καλωσορίζω λοιπόν δύο εκπροσώπους από τις κάτω χώρες, από το Ίδρυμα Βαρθολομαίου. Αν θέλετε είναι από τα παγκόσμια κέντρα αυτό ένα που ε, αξιολογούν αυτό το θέμα. Είναι ο Μάρτιν Χάουτεπεν και ο Έρικ Φέρμαν από τις κάτω χώρες που συντονίζουν την παρουσίαση. to welcome. Και επίσης να καλωσορίσω την ε, κυρία Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου που ηγείται σε μια σχολή ε, ε, από σκυλιά οδηγούς τυφλών και μας δείχνει πόσο δύσκολο είναι και ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Και επίσης να καλωσορίσω ε, το ε, και από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Εργάζεται πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το θέμα και συμφωνώ μαζί του. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Ευρώπη έχουμε καθυστερήσει σε σύγκριση ε, με κάποια κρατημέλη και τον κόσμο ολόκληρο. Αν μου επιτρέπετε τώρα να δώσω το λόγο στους δύο Ολλανδούς ε, εμπειρογνώμονες. Fine. Good. Yes. So, thank you very much. Happy to give you the floor. And your slides will come up here and on the last screen. Εδώ θα βγουν οι διαφανίες σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρουσιάσω μερικά ε, παραδείγματα. Το πρώτο θέμα για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων Βλέπετε εδώ ορισμένα στοιχεία που τα πήρα από μία παρουσίαση πριν από μερικού μήνε. δεν αφορά μόνο του ανθρώπου με αναπηρίε, αφορούν και του ανθρώπου ε, που μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα λόγω της συγχωρήπανση, λόγω του εξωτερικού φωτός, ε, ε, μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα οδηγώντα το αυτοκίνητό του ή τα μάτια που γυράσκουν και δυσκολεύονται πούμε, να διαβάσουν ε, τα email τους. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, προβλήματα. Μπορεί να έχει κανείς κάποιες κινητικές ε, δυσκολίες, αλλά όλος ο κόσμος το έχει αυτό αν έχει πάρα πολλές λακκούβες ο δρόμος, για παράδειγμα, ή όταν διαβάζει κάτι σε ένα μικρό τάμπλετ. Η προσβασιμότητα λοιπόν αφορά όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως ε, του αν είναι κάποιος άτομο με αναπηρία ή όχι. Συμπεριλαμβάνονται αυτοί με αναπηρίες και άνθρωποι που έχουν κάποιους περιορισμούς ή κάποιοι που έχουν προσωρινές αναπηρίες. Οι μηχανές αναζήτησης θέλει κανείς να μπορεί να, βρίσκεται, να το βρίσκει κανείς στο ίντερνετ ε, ξέρετε ότι είναι ε, τυφλό και εν μέρη κουφό ε, το παγκόσμιο συστός, οπότε αν θέλει κανείς κάποιος να μπορεί να αναζητηθεί ε, στο ίντερνετ πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Ε, το 80 με 90% βέβαια ε, το κάνουν ήδη αυτό. 4,5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού κάτω των 65 έχει προβλήματα οράσεως και ένας στους 5 έχει αχρωματοψία. Ε, η επικουρική τεχνολογία τα κάνει όλα. Δεν χρειάζεται κανεί να έχει ειδικού ιστότοπου. Αν κάποιο ε, ε, είναι σχεδιαστή, χρειάζεται απλώ τι προδιαγραφέ, όπω για παράδειγμα ένας ε, σωστό μπογιατζής χρησιμοποιεί τη σωστή μπογιά για να βάψει το σπίτι του, αναλόγω με το αν θέλει να το βάψει από μέσα ή, από έξω. Ε, υπάρχουν επίσης ορισμένα στοιχεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αν κάποιος ε, ε, επιμελείται του περιεχομένου, χρειάζεται κάποια εκπαίδευση αν υπάρχει ένα ελληνικό κείμενο για παράδειγμα και ξαφνικά είναι, γίνεται αγγλικό, θα πρέπει να αλλάζει η φωνή που ακούγεται από τον υπολογιστή, ε, ώστε να μην ακούγονται τα αγγλικά με ε, ελληνική προφορά, εκτός αν σε κάποιον αρέσει αυτό βεβαίως. Ε, δεν χρειάζεται να κάνει κανείς τίποτε το ιδιαίτερο εκτός από το να χρησιμοποιήσει τους, ε, τις προδιαγραφές ε, για να υπάρχει μεγέθυνση της γραμματοσυράς ή για παράδειγμα αν χρησιμοποιεί κανείς τεχνολογίες αφής ή αναγνώρισης φωνής αν είναι κανείς επιμελητής περιεχομένου, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία για να κάνει τη δουλειά του σωστά. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι οι οποίοι έχουν, προ... έχουν σωματικές αναπηρίες. 6,4% ε, των ε, Ευρωπαίων ε, έχουν προβλήματα χρήσης των χεριών τους Ευρω... μερικοί ευρωπαϊκοί στο οποίο έχουν πολύ μεγάλα μενού και αν χρησιμοποιεί κανείς το tab για να πάει από item σε item, μερικές φορές πρέπει 40 ε, με 50 φορές να πατήσει το tab για να φτάσει εκεί που θέλει. Και αν κάνει κάποιος την επιλογή πρέπει να ε, πατήσει τόσες φορές το κουμπί ξανά ο μόνος τρόπος να το παρακάμψει κανείς αυτό είναι να υπάρχει το skip link, ένας σύντομος ε, σύνδεσμος πάνω-πάνω στη σελίδα. Οι περισσότεροι ιστότοποι το έχουν αυτό, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα τα προβλήματα ΚΟΗ, 3,1% ε, κάτω των 65 έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ε, τα προβλήματά τους είναι λοιπόν οπτικοακουστικό υλικό χωρίς ε, υπότιτλους ή χωρίς κείμενο. Αν κάποιος ας πούμε θέλει να δείξει ένα βίντεο σε κάποιο εστιατόριο που υπάρχει θόρυβος ή κάθεσε σε ένα μπαρ και θέλει να ακούσει ένα ειδησιογραφικό πρόγραμμα, ξέρετε ότι πρέπει να βάλετε τον ήχο πολύ πιο δυνατά εκτός εάν ε, υπάρχουν ε, υπότιτλοι. Το πρόβλημα με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής ε, είναι η νοηματική. Ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός. από, βέβαια, εντάξει, οι υπότιτλοι ε, ε, εξακολουθούν να αποτελούν μια καλή τεχνολογία και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, οι επίκτητες αναπηρίες, ε, όπως για παράδειγμα αυτισμός, δυσλεξία, προβλήματα ανάγνωσης, ADHD, αφασία... Αυτό όμως ε, δεν αποτελεί μόνο μία, ε, ένα τεχνικό ζήτημα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι άνω των 65 ε, που έχουν, αντιμετωπίζουν, έχουν κάποιες αναπηρίες όσο μεγαλώνουν. η, οι άνθρωποι άνω των 65 είναι όλο και αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού μας. Δεν ε, έχουν τις αναπηρίες ε, που γνωρίζουμε εμείς, αλλά έχουν κάποια προβλήματα ακοής, ε, προβλήματα οράσεως. Το να είναι ο ιστότοπος λοιπόν πιο προσβάσιμος, γενικά θα είναι πιο προσβάσιμος και για εκείνους. Τώρα, οι περιορισμοί ε, που ανέφερα προηγουμένως, ε, το φως, ε, ο ήλιος, το να μην έχει κανείς τα τελευταία plug-in, το να χρησιμοποιεί ένα iPad, θα γνωρίζετε ότι όταν πηγαίνει κανείς σε έναν ιστότοπο χρειάζεται plug-ins τα οποία δεν υποστηρίζονται από το iPad Ε, ξέρετε ότι για πολλά τάμπλετ ισχύει αυτό. Αν δεν υποστηρίζεται, αν η τεχνολογία των plug δεν υποστηρίζεται, θα πρέπει κάποιο να αντιπαρέλθει κάπως αυτό το πρόβλημα. Οι διάφορες τώρα συσκευές, ε, το συζητήσαμε μόλις αυτό, το ανέφερα μόλις αυτό, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν δουλεύουν, ε, πάνω, δεν δουλεύουν στο iPhone. Γνωρίζετε ότι τα iPhone, τα iPad, τα Android ε, τηλέφωνα και οι τα tablets Android έχουν κάποια θέματα προσβασιμότητας. Η προσβασιμότητα είναι πολύ καλή, όμως για παράδειγμα, πολλοί τυφλοί χρησιμοποιούν ε, το iPhone γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πολλά πράγματα μέσω της φωνής. Ε, μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να διαβάσουν SMS, ε, να χρησιμοποιήσουν τα πάντα στο iPhone τους στο τηλέφωνό τους. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί ιστότοποι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία το αναφέρει ήδη σε συνολικά πάνω από ένα εκατομμύριο ε, ηλεκτρονική, ε, ιστότοποι ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ένα μικρό ποσοστό μόνο είναι προσβάσιμο. Και εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον στις κάτω χώρες, 10% λιγότερο από 10% είναι προσβάσιμα, προσβάσιμοι ιστότοποι δημόσιοι ιστότοποι, είναι... Ε, υπάρχει κάποια βελτίωση, αλλά σε μικρό ποσοστό κατ' έτος. Αν δει κανείς την αγορά για την προσβασιμότητα του ιστότοπου, υπάρχει το πρόβλημα της εναρμόνισης. Υπάρχουν ε, τοπικοί υπολογισμοί, μέθοδοι υπολογισμού της ε, προσβασιμότητας και υπάρχει ένας κίνδυνος κατακαιρματισμού. Επίσης, για το κλάδο υπάρχει μια ανάγκη εναρμόνιση. Ε, φανταστείτε ότι είστε μια χώρα, ότι είστε μια εταιρεία που δεν δουλεύει μόνο στην Ολλανδία ή στο Βέλγιο, αλλά σε 20 χώρες. Θα χαρεί, θα χαρεί πάρα πολύ με μια, με, με μια κατευθυντήρια γραμμή που χρησιμοποιείται παντού και που υπολογίζεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Η συμβατότητα Μερικά παραδείγματα. Ένα απλό παράδειγμα. Το κείμενο ALT είναι ίσως ε, πολύ τεχνικός όρος, αλλά είναι τέλο πάντων σύντομη περιγραφή του τι σημαίνει ένας ε, όρος. Δηλαδή, ε, το YouTube έχει ως ALT κείμενο το logo, logo YouTube. Αυτό θα διάβαζε το website σε κάποιον που είναι τυφλός. YouTube, logo YouTube τα φινλανδικά μου δεν είναι πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα από τη φινλανδική κυβέρνηση. Είναι η δικτυακή πύλη της φινλανδικής κυβέρνησης. Ε, το λόγο είναι, είναι το μοναδικό πρόγραμμα που λέει τι ακριβώς ε, είναι αυτό το, ε, αυτός ο ιστότοπος. Αν δεν σας το διαβάσει κανείς, δεν καταλαβαίνετε τίποτε. Πρέπει να διαβάσει κανείς και το υπόλοιπο κείμενο. το fix θα γίνει όμως σε τρία δευτερόλεπτα. Απλώς προστίθεται το alt Δεν είναι κάτι λοιπόν που θα σας, ε, ε, θα, θα, θα χρειαστείτε μέρες για να το κάνετε. Είναι κάτι το οποίο μπορείτε να διορθώσετε σε, τρεις, ε, σε τρία δευτερόλεπτα. Τώρα το πρόβλημα της συνέπειας. Αν δει κανείς έναν ιστότοπο, είναι καλό όσοι έχουν επίκτητες αναπηρίες να έχουν μια συνεπή πλοήγηση στο ίντερνετ. Βλέπετε ας πούμε στα αριστερά ένα μενού και στην επόμενη σελίδα δεν βλέπετε μόνο ένα μενού στα αριστερά, αλλά είναι και, υπάρχει και ένα μενού ε, στο πάνω μέρος της σελίδας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει στις κατευθυντήριες γραμμές, η συνέπεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα σας πάρει 5 λεπτά για να το διορθώσετε. Τώρα τα βίντεο χωρίς ε, υποτιτλισμό για ε, τους βαρύκοους ή τους τυφλούς. Εδώ βλέπετε ας πούμε ένα νηστότοπο του Λουξεμβούργου 20 δευτερόλεπτα έχει το βίντεο, ε, είναι το βίντεο και νομίζω ότι θα χρειαστεί επιδιόρθωση, δηλαδή προσθήκη ε, υποτίτλων, δύο λεπτά. Ένα ε, παράδειγμα τώρα από έναν ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ υπάρχει ένα βίντεο και το βίντεο έχει, όπως μπορεί να μπορείτε και να δείτε, είναι πολύ μικρά τα γράμματα, υπάρχουν υπότιτλοι. Και μπορεί μάλιστα να διαλέξει κανείς από 20 ή παραπάνω διαφορετικές γλώσσες, να αλλάξει κανείς τον υποτιτλισμό σε ό,τι γλώσσα επιθυμεί. Έτσι θα έπρεπε λοιπόν να είναι τα βίντεο. Ένα ακόμη παράδειγμα ε, του ιστότοπου εσόδων ε, της Ιρλανδίας. Έχει φλάσο αυτό το, ε, το βίντεο και ξέρετε ότι το iPad δεν έχει υποστήριξη flash, οπότε ε, αν το βλέπει κανείς από το iPad δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτε με τους ε, φόρους του, κάτι το οποίο τέλος πάντων κατά τη γνώμη μου δεν είναι κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, επίσης δεν μπορεί κανείς να έχει ε, υπηρεσίες πληκτρολογίου σε Chrome, ε, ούτε καν στους υπολογιστές ε, Mac με λειτουργικό OS X. Αυτά λοιπόν η σύντομη παρουσίασή μου. Good. Uh, thank you very much. So... Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Εσύ θα έχεις τώρα το γενικό πρόσταγμα, Γιώργο, εσύ διευθύνεις τη συζήτηση, πες μας τώρα. Ε, τώρα είδαμε τις τεχνικές ε, προδιαγραφές και απαιτήσει. υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές και είναι πάρα πολύ εύκολο να ε, ε, ακολουθήσει κανείς τις οδηγίες. Δεν είναι τίποτα το μαγικό, απλή τεχνολογία είναι. Να ακούσουμε τώρα την κυρία Γκέρτσου, η οποία θα μας δείξει πώς ε, βλέπει μια ιστοσελίδα, έναν ιστότοπο και κατά τύχη είναι η δική μου ε, του Ευρωβουλευτού και η κυρία Γκέρτσου θα μας ε, παρουσιάσει και θα μας περιγράψει τι μπορεί να αντιληφθεί από τον ιστότοπο αυτό ε, τυφλή. Um, my name is Maria. Καλημέρα σας. Λέγομαι Ιώνα Μαρία Γκέρτσου. Ίδρυσα μία σχολή ε, σκύλων οδηγών τυφλών ε, στην Ελλάδα ε, στο παρελθόν. Ήμουν ειδική στο Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα για θέματα πρόσβασης και πρέπει να σας ε, εξηγήσω τώρα πώς μπορεί κάποιο άτομο που έχει πρόβλημα όρεσης, είναι τυφλό όπως εγώ, ε, να χρησιμοποιήσει και να επισκεφθεί έναν ιστότοπο όπως του κυρίου Χατζή Μαρκάκη. Επιλέξαμε αυτόν τον ιστότοπο και ο ίδιος να το ε, έχει στη διάθεση και να είναι πλήρως προσβάσιμος για ανθρώπους με αναπηρίες. Είμαι εδώ με την ομάδα μου ε, εκπροσωπούμε την Ελλάδα και με τον κύριο Ιωάννη Μπασδέκη που ε, είναι και ο προγραμματιστής ε, αυτού του ιστοτόπου και το προγραμμάτισε ακριβώς για να είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες. Για να συγκρίνουμε λοιπόν δύο ιστοτόπους τώρα. Είναι λίγο πρωτόγονος ο τρόπος με τον οποίο διαβάζω το ε, κείμενο. Δεν έχω μεγάλο προϋπολογισμό και κατέβασα από το διαδίκτυο ε, δωρεάν ένα λογισμικό freeware. Να σας δείξω πρώτα την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του κυρίου Χατζημαρκάκη που δεν είναι προσβάσιμη για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Ζητώ συγγνώμη. το πρόβλημα που έχουμε και με την οθόνη ανάγνωσης είναι ότι δεν είναι συχνά ε, συμβατά τα συστήματα αυτά με άλλους υπολογιστές και θα πρέπει να το προσαρμόσω. Λοιπόν, εδώ έχουμε την παλιά ιστοσελίδα του κυρίου Χατζη Θα προσπαθήσω να το διαβάσω. Αλλά εγώ δεν ξέρω που βρίσκομαι τώρα στην οθόνη. Γιατί δεν έχει ε, προγραμματιστεί για να χρησιμοποιείται με βοήθεια ανάγνωσης και ε, χωρίς ποντίκι. Προσπαθώ λοιπόν να προσανατολιστώ πάνω στην οθόνη αυτή, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα ε, η οθόνη μου περνάει από σύνδεσμο σε σύνδεσμο από μόνη της και εγώ δεν ξέρω ακριβώς που βρίσκομαι. Yeah, I um, a bit when when we're nervous we lose the simple things. <laughs> Λοιπόν, ε, είναι αυτή λοιπόν λέγαμε μια ιστοσελίδα που δεν έχει χάρτη οδηγίες χρήσεως για τους ανθρώπους με αναπηρίες δεν έχουμε shortcuts δηλαδή για να μπορούμε γρήγορα να περνούμε ας πούμε, στη βασική σελίδα, στην αρχική σελίδα ή ε, σε άλλα σημεία του ιστοτόπου. Είναι πάρα πολύ διάχυτη η πληροφόρηση ώστε κάποιος ε, τυφλός ή με προβλήματα όρασης δεν μπορεί να πλοηγηθεί. Um, the, uh, Λοιπόν, διαβάζει το υπολογιστή στην ε, πληροφόρηση, αλλά είναι διάχυτη και τα διάφορα link ε, ε, είναι κάτι που μας οδηγεί σε σύγχυση. Αν δούμε λοιπόν πώς έχει η νέα σελίδα, που είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες, So, Λοιπόν, αυτή είναι η νέα μορφή. Ε, τώρα βρίσκομαι στην ε, βασική αρχική σελίδα ε, και οθόνη και θα προσπαθήσω να σας δείξω πώς είναι η πλοήγηση. Μου μιλάει ο αναγνώστης της οθόνης. Έχω ένα πρόβλημα γιατί ο υπολογιστής μου είναι στα ελληνικά και ο αναγνώστη οθόνη διαβάζει τα αγγλικά. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ε, ζωή. Ε, θα αλλάξω λοιπόν τη γλώσσα για να διαβάζει την ιστοσελίδα στα αγγλικά, αλλά συγκρούεται με τα ελληνικά Windows πλέον. okay. So this is the main page of uh, Mr. Georgos Και πάλι αυτή είναι η αρχική σελίδα, βασική σελίδα του τόπο ε, ιστοτόπου του κύριου Χατζημαρκάκη.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 με βοηθήσει για να βρω τα βασικά settings ε, προσβασιμότητας. Τις βασικές ρυθμίσεις λοιπόν. So στο βασικό μενού τώρα της προσβασιμότητας. Και αντί λοιπόν για πλοήγηση δεξιά και αριστερά και τυχαία στην ιστοσελίδα και επειδή δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ποντίκι, χρησιμοποιώ το πληκτρολόγιο. Με έχει ενημερώσει ήδη το σύστημα ότι αυτό μπορώ να το κάνω και ε, μεταφέρθηκα αμέσως ε, στις ρυθμίσεις προσβασιμότητας ε, του ιστοτόπου αυτού. Και τώρα με ενημερώνει ο υπολογιστής ότι μπορώ να πατήσω ένα πλήκτρο και να πάω κατευθείαν στο σύνδεσμο που με ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνω με το πληκτρολόγιο στον ιστότοπο. Και να διατρέξω όλες τις πληροφορίες μέχρι να καταλάβω πού ακριβώς βρίσκομαι στην οθόνη. Επιστρέφουμε στην αρχική σελίδα και πίεσα ένα σύνδεσμο για να γυρίσω ε, στην ε, αρχική σελίδα και τώρα ε, με οδηγεί αυτό το σύστημα να διαβάσω τα διάφορα άρθρα. Technology is not very uh, well δεν μας βοηθάει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Η τεχνολογία δεν είναι το πλευρό στο πλευρό μας. Τα σκυλιά είναι πιο αξιόπιστα. So now I try to navigate in the website. Τώρα προσπαθώ να πλοηγηθώ λοιπόν στην ιστοσελίδα και να ανατρέξω σε κάποιο θέμα που θα με ενδιαφέρει. Με ενημερώνει το σύστημα για τους συνδέσμους που έχω και μπορώ να πατήσω το πλήκτρο press και να ε, βρεθώ εκεί ακριβώς που θέλω για ε, διάφορες ε, ενημερώσεις ανακοινώσεις τύπου, δελτία τύπου. Και μπορώ έτσι να δω τι ανακοινώσεις, τι δελτία τύπου μπορώ να ακούσω. Να σας δείξω και μια άλλη ρύθμιση, αν μπορώ, αν τα καταφέρω. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Okay. Um, so Αυτά. Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα. Καταλάβατε, φαντάζομαι. Πώς μπορεί κάποιος με προβλήματα όρεσης και τυφλός να χειριστεί αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Χατζημαρκάκης και για μένα αυτό ήταν πραγματική επίδειξη. Um, for first time Για πρώτη φορά Ε, βλέπω να μου το εξηγεί κάποιος που είναι ο αποδέκτης και ο χρήστης. Γιατί οι περισσότεροι έχουμε διαφορετική προσέγγιση σε κάθε ιστότοπο. Και βλέπετε και οι ίδιοι πόσο δύσκολο είναι στην πράξη να χρησιμοποιήσει κανείς ένα τέτοιο σύστημα και πόσο χρόνο χρειάζεται κανείς. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε επιγόντως κάποια απλούστευση, νόμοθεσία, εναρμόνιση στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη για να χρησιμοποιούμε αυτά τα συστήματα. Γκέρτσου ήρθε από την Ελλάδα και την ευχαριστώ που ήρθε για να μας τα δείξει αυτά. Και αυτό αφορά 15% του πληθυσμού στην Ευρώπη. Βλέπετε λοιπόν το πρώτο αυτό εμπόδιο είναι τεράστιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρτσου και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον Ροδόλφο Κατάνη, τον επόμενο μιλητή, να λάβει το λόγο. Εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you. Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, είδατε τις δυνατότητες, είδατε τις δυσκολίες. Νομίζω πως αρχίζετε να καταλαβαίνετε πως η αλλαγή είναι δυνατόν να γίνει. Θα πρέπει έχει υπάρξει μια ιστορική μετακίνηση από το υλικό στο άϊλο όσον αφορά την παγκόσμια, το παγκόσμιο περιβάλλον επικοινωνίας. Η προσβασιμότητα είναι σημαντική για την παιδεία, για την αποκατάσταση, για την κοινωνική ζωή, για την πολιτιστική ζωή και για την πολιτική ζωή βεβαίως. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους οργανισμούς, διοικητικούς οργανισμούς και ούτω καθεξής, καθίστανται όλο ένα και πιο πρακτικοί και απλοί για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Εμείς σίγουρα χρειάζεται να έχουμε μια προσέγγιση ε, με επίκεντρο το χρήστη. Νομίζω πως είναι σαφές τώρα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται εγώ να το πω ότι κάτι δεν πάει καλά όσον αφορά την προσβασιμότητα. Οι μελέτες της Κομισιόν δείχνουν πως μόνο και το 10% ή μάλλον λιγότερο από το 10% των δημοσίων ιστοτόπων είναι προσβάσιμα. Το μίμηση αυτού του ποσοστού ε, ισχύει για τους ιδιωτικούς ιστότοπους. Θα πρέπει να σας πω το εξής. Υπάρχει οικονομική προοπτική εδώ, διότι η προσβασιμότητα μπορεί να δώσει όθηση, όθηση στις μικρομεσαίες, που είναι η πιο σημαντική παραγωγή προσβάσιμων ε, ιστοτόπων δεν είναι δαπανηρό κάτι τέτοιο. Είναι μια ευκαιρία, δεν είναι μια δυσκολία. Αλλά δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι το να αποκλείεται κανείς, το να μπαίνει στην άκρη στην κοινωνία, είναι απαράδεκτο για τόσο πολύ κόσμο. Όχι μόνο ανθρώπους με Είδαμε πως είναι πρόβλημα και για τους ε, ηλικιωμένους και για τους λιγότερο ε, μορφωμένους που χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Νομίζω πως είναι σημαντικό, είναι μάλιστα ουσιώδης το να κατανοήσουμε πως η πρόταση αυτή είναι ανεπαρκής είναι και πολύ αργά, γιατί αν χρειάζεται χρόνος θα πρέπει να δώσουμε χρόνο. Αλλά είναι λιγοστά αυτά που προτείνονται. Μόνο 12 κατηγορίες προβλέπονται και μάλλον ε, αναγνωρίζονται που χρονολογούνται από το 2001. Πάνω από 10 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Μέχρι το 2015 θα έχουμε τεράστια αύξηση της ανάγκης προσβασιμότητας. Και πλέον ήγηκε και η ώρα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ε, μετατρέψουν όλα αυτά σε πραγματικότητα. Δυστυχώς τον επόμενο χρόνο θα υπάρξει πλήρης αλλαγή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα έχουμε νέο κοινοβούλιο, νέα επιτροπή και πραγματικά θα θέλαμε <clears throat> να περάσει αυτό το νομοθέτημα πριν να γίνουν όλα αυτά τον επόμενο χρόνο, πριν τον Ιούνιο, δηλαδή του 2014, όταν θα λήξει αυτή η θητεία. Θέλουμε να ολοκληρωθεί ένα φιλόδοξο νομοθέτημα σύμφωνα με την ε, λίγη αναμενόμενη πράξη περί προσβασιμότητας, την οριζόντια οδηγία περί μη ε, διακρίσεων, που κάπου και αυτή λαγοκοιμάται, Υπάρχουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικέ ανάγκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε πω οι ανάγκε του θα ληφθούν υπόψη και θα γίνουν σεβαστέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Grazie ε, ευχαριστώ πολύ, Ροδόλφο. Ε, ολοκληρώνεται έτσι η παρουσίαση. Θα έχουμε και μια πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση από τον συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Οικονομικό και Κοινωνικό ε, Συμβούλιο, Επιτροπή ε, δηλαδή, που ζητήσαμε τον κύριο Πιέρ Άμπελκαρ που και εκείνος έχει πρόβλημα όρασης και θα κάνει μια πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση για την έκθεσή του που αποτελεί μια πολύ καλή βάση για μας. Και έτσι ολοκληρώνεται η παρουσίαση Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πολύ που τα διοργάνωσες όλα αυτά. Εγώ λοιπόν προτείνω, εφόσον έχουμε εδώ τους καλεσμένους μας, να δούμε και την παρουσίαση του κ. Μπινγκάλλα, αν συμφωνείτε κι εσείς. Διότι θα έχουμε έτσι την ευκαιρία ε, εμείς ε, ε, να το συζητήσουμε μαζί με τους Σκιώδης και αργότερα. Ενώ τώρα καλύτερα είναι να έχουμε μια πλήρη ανταλλαγή απόψεων και να εκμεταλλευτούμε την παρουσία των προσκεκλημένων μας. Και θα, έχω για την θα δώσω το λόγο και στην Κομισιόν, αν συμφωνείτε κύριε Χατζημαρκάκη. Λοιπόν, πιστεύω πως θα ήταν καλύτερη ιδέα να ακούσουμε την, την, άλλη, την επόμενη παρουσίαση. Πού βρίσκεστε, μπορείτε να κάνετε την παρουσίασή σας ήδη, είστε έτοιμος. και μετά θα ελέγξουμε το χρόνο για να δούμε αν πρέπει να προβούμε στις τελικές παρατηρήσεις και να συνεχίσουμε και τη συζήτηση αργότερα. Πολύ τιμή συζήτηση σήμερα. Κύριε Σαβίγκα, λοιπόν, από την ΟΚΕ, με τα χαράς σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο γιατί είμαι και εγώ περίεργος να ακούσω τις απόψεις ε, που θα εκφραστούν εδώ στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ καταρχήν πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε για να παρουσιάσω την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, την φωνή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, εργοδοτών, εργαζομένων και πολλών ενδιαφερομένων και ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αρχική γνωμοδότηση, αλλά στην Επιτροπή μας υπάρχει ευρεία συνένεση για τα όσα θα σας πω εγώ σήμερα και όπως είπα θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, οπότε θα περάσω αμέσως στο πιο ουσιαστικά σημεία. Έχω το προνόμιο κάποιοι από τους προηγούμενους ε, μελετές να έχουν παρουσιάσει το θέμα και να σας έχουν δώσει μάλιστα και κάποια αριθματικά στοιχεία καθώς και πολύ πρακτικά σας εξήγησαν πώς λειτουργεί η προσβασιμότητα ή δεν λειτουργεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορώ να σας πω για λογαριασμό μου ότι ε, χρησιμοποιώ του υπολογιστέ καθημερινά. Ποτέ δεν χρησιμοποιώ το ποδίκι γιατί δεν είναι δυνατό να το κάνει κανεί ω ε, τυφλό. Ε, πέρα από την προσωπική μου εμπειρία, οι απόψει τη. ΟΚ τώρα. Συμφωνούμε με τον κύριο Κατάνη ότι θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το θέμα της επέκτασης ε, του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ώστε σταδιακά να καλύψει όλους ε, τους ιστότοπους των δημοσίων οργανισμών και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω το γιατί. Η φιλοδοξία μας, και νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτό, ε, είναι ότι η προσβασιμότητα θα πρέπει να είναι ένα αυτόματο κομμάτι της διαδικασίας κατασκευής ενός ιστοτόπου είτε της ε, παρουσίασης περιεχομένου ε, στο δίκτυο αν είσαι δημόσιος Θα πρέπει αυτό λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι μια αυτόματη, ε, ένας αυτόματος κρίκος της αλυσίδας στη διαδικασία κατασκευής ενός ιστοτόπου. Θα πρέπει να είναι μέσα στο software που χρησιμοποιούν οι συντάκτες των ιστοτόπων ώστε να και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και γι' αυτό και δεν αρκεί δεν αρκούν οι προδιαγραφές του καταλόγου του 2001 που είναι ήδη ξεπερασμένος, πεπαλαιωμένος όπως είπε και ο κύριος Κατάνη. Εφόσον θέλουμε λοιπόν, εφόσον, αν μάλλον επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή, θα δημιουργήσουμε αυτή την κρίσιμη μάζα που θα κάνει τους φορείς της αγοράς στο, στην αγορά προσβασιμότητα να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα ίδια στάνταρ. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως τα στάνταρ τα οποία, για τα οποία εμεί μιλάμε τώρα στις προτάσεις για οδηγίας είναι στάνταρ προδιαγραφές που διευκρινίζονται σε διεθνές επίπεδο. Είναι οι κατευθυντήριες γραμμές 2.0 που ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο για την προσβασιμότητα. Εάν δηλαδή παραμένουμε σε αυτές τις προδιαγραφές θα μπορούμε να προσφέρουμε προσβασιμότητα στους ιστοτόπους ε, για, στην παγκόσμια αγορά. Αυτά λοιπόν για το πεδίο εφαρμογή. Είναι σημαντικό δε νομίζω να πούμε ότι δεν είναι αυτόματο μόνο επειδή κάποιο ιστότοποι δημοσίων οργανισμών τηρούν τις ε, προδιαγραφές προσβασιμότητας, το κάνουν όλοι. Σε κάποια κράτη-μέλη Υπάρχουν απαιτήσει ε, προσβασιμότητας για κάποιους ιστότοπους, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ε, περνά αυτόματα και στους υπόλοιπους ιστότοπους. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς και συνεπείς απαιτήσει σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, γιατί αυτό διευκολύνει και την εφαρμογή Τώρα, τα συμπληρωματικά παράπλευρα μέτρα που θα θέλαμε να προτείνουμε και που θα είναι και το τέλος της δικής μου παρουσίασης. Αυτό που προτείνουμε είναι να πούμε ότι πέρα από τον μηχανισμό παρακολούθησης θα πρέπει να υπάρχει και διευκόλυνση για τους πολίτες να αναφέρουν την, προσβασιμότητα ή μη των ε, ιστοτόπων, ώστε ένας απλός τρόπος ώστε οι πολίτες να μπορούν να στείλουν ένα mail με, μια, ένα σύνδεσμο, ένα link για το προσβάσιμο ή μη προσβάσιμο ιστότοπο στο αρμόδιο όργανο έτσι ώστε ε, πολύ εύκολο τρόπο να μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας και τα κράτη-μέλη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές στη σύστημα αναφοράς τους για την παρακολούθηση των οδηγιών. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τις εμπειρίες των χρηστών με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε για το crowdsourcing, δηλαδή την απορρόφηση, ε, την χρήση μάλλον του κόσμου για να μπορούμε να λειτουργούμε σε διάφορα επίπεδα. Έτσι λοιπόν να μπορέσουμε να δουλέψουμε και με ιστοτόπους, που, με, μάλλον με εταιρείε που ενημερώνουν τους ιστοτόπους ε, για να τους ενημερώσουμε και οι κοινωνική εταίροι θα πρέπει σίγουρα να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Να υπογραμμίσω κιόλας ότι συζητάμε πολύ τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και πώς αυτές θα ληφθούν υπόψη. Και αυτό που λοιπόν που λέμε καταρχήν είναι ότι οι κινητές εκδοχές των ιστοτόπων θα πρέπει να καλύπτονται ρητά από την οδηγία ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα είναι, θα είναι ασφαλής και για το μέλλον Από πρακτική άποψη δεν είναι πρόβλημα, γιατί αυτό περιλαμβάνεται στις τις διεθνεί προδιαγραφέ προσβασιμότητα. Επίση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολλά σώματα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν ε, εφαρμογέ και για τα smartphones και για τι ταμπλέτε, ε, για να δίνουν τις πληροφορίες στους πολίτες και εν πάση περιπτώσει αυτά τα apps οι εφαρμογές ενσωματώνονται στη λειτουργία των ιστοτόπων των δημοσίων οργανισμών. Οπότε στο βαθμό που αυτό είναι νομικά δυνατόν, η παροχή αυτών των εφαρμογών στους πολίτες θα πρέπει να καλύπτεται επίσης στο βαθμό που είναι ενσωματωμένο στις λειτουργίες ε, του ιστοτόπου των δημοσίων αυτών οργανισμών. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, της Κομισιόν, και έπρεπε ήδη να έχει γίνει ε, αλλά ανησυχούμε όσον αφορά την καταλληλότητα του πεδίου εφαρμογή. Το πιστεύω ότι θα πρέπει να επεκταθεί και ότι με σαφή τρόπο να αναγκάσουμε τον κατακαιρματισμό αυτών που επικρατεί στην ενιαία αγορά αυτή τη στιγμή να τον ε, ξεπεράσουμε και να βρούμε και κατάλληλου τρόπους για να το κάνουμε αυτό. Αυτά για την ώρα. Πολύ ευχαρίστω να προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις σας και να προσβλέπω στη συνέχιση του διαλόγου με τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας μέχρι στιγμής. Uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ε, σαφείς ε, επεξηγήσεις. Μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για το δικό σας χρονοδιάγραμμα. Ε, πότε θα εγκριθεί η δική σας έκθεση από την ΕΟΚΕ, στις 22 Μαΐου. Ωραία. Δυστυχώς δεν θα έχουμε συζήτηση, δεν θα έχουμε χρόνο για περαιτέρω συζήτηση σήμερα, αλλά ευχαρίστω να σας καλέσουμε στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων. Πρέπει να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χατζημαρκάκη, γιατί έχουμε και πολλές ψηφοφορίες στις 10 η ώρα και έχουμε περιορισμένο χρόνο συνεδρίασης. Ήταν πάντως πάρα πολύ χρήσιμο το, τα στοιχεία αυτά που λάβαμε. Να δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Χατζημαρκάκη για να αποφασίσει αν θέλει να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια για το πώς θέλει να συνεχίσουμε. Θέλετε να ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον. Κύριος Χατζημαρκάκης, επειδή θα ψηφίσουμε, κανονικά ψηφίζουμε στις 10 ε, παρα 5, ας, μας, ε, ας ακούσουμε τον κύριο Ιακωβίδη κάποια άλλη στιγμή, αν δεν τον πειράζει πολύ, να μου δώσετε τη δυνατότητα ίσως κύριε Πρόεδρε μετά από την ψηφοφορία να ε, πάρω το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Απιτκάρτ ε, ε, που είναι ο εισηγητής του θέματος αυτού. Ε, πάρα πολύ συνοπτικά μας παρουσίασε τις σημαντικότερες πτυχές αυτής της νομοθεσίας και χαίρομαι που και εσείς στην ΟΚΕ υποστηρίζετε σε γενικές γραμμές αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε όμως πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη για να το απλοποιήσουμε. Για να την απλοποιήσουμε θα το κάνουμε μαζί. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά σας ως βάση για μας, για το Κοινοβούλιο. Από τη στιγμή που εσείς μια και ζείτε το πρόβλημα, ε, είστε πολύ πιο ε, κατάλληλος ε, εισηγητής. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ε, ολοκληρώσω εδώ κύριε Πρόεδρε και να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ναι, δεν θα έχουμε χρόνο όμως λέει ο Πρόεδρος ε, να το συζητήσουμε μετά την ψηφοφορία. Ε, προτείνω μία δεύτερη ανταλλαγή απόψεων με εσά και με τους σκιώδεις εισηγητές. και 17 και 10, με 19 Μαΐου θα, συγγνώμη, Ιουνίου θα ε, συζητούσαμε κανονικά την, ε, θα, θα ψηφίζαμε την γνωμοδότησή σας, οπότε νομίζω ότι στις 7 ε, Μαΐου μπορούμε να έχουμε μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Στις 22 Μαΐου θα στείλουμε τότε σε μετάφραση την, την έκθεσή σας, οπότε θα έχουμε το χρόνο μέχρι τις 17 Ιουνίου. Ήθελα να σας πω ότι μεταδίδονται οι συνεδριάσεις μας στο διαδίκτυο, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια είναι προσβάσιμος ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και δεν ξέρω ίσως ο κύριος Χατζημαρκάκης και οι σκιώδες συζητητές θέλουν να, σώσουν, να, να, να θέσουν αυτό το ζήτημα ε, κατά πόσο δηλαδή μπορούν ε, ε, οι άνθρωποι με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση και να, αλληλο, να αλληλεπιδρούν με, τους, με τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως, ε, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ από την πλευρά μου για να μπορέσετε να το συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας. Ξέρω, κύριε Χατζημαρκάκη, ότι θα το λάβετε υπόψη, γιατί πραγματικά είναι μία, ε, μια πολύ, ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ υποδειγματική έκθεση, γιατί πρέπει εμείς πρώτοι να κάνουμε προσβάσιμο τους ιστότοπους μας. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα και εσάς ως συζητητή, αλλά και τους κοιόδης συζητητές. Να ολοκληρώσω λοιπόν λέγοντας πόσο ευγνώμονες είμαστε σε όλους όσους ήρθαν σήμερα να υποστηρίξουν τις εργασίες μας και βεβαίως ε, και η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο, το λέω αυτό για όσους παρακολουθούν. Έχουμε επίσης και ένα newsletter, ένα ενημερωτικό φυλάδιο, αν θέλετε, ε, μπορείτε να λάβετε γνώση και έχει μάλιστα και links ε, στα οποία μπορείτε να ε, πάτε για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τις εργασίες μας και ε, όταν το σχέδιο εκθέσεως του κυρίου Χατζημαρκάκη θα είναι διαθέσιμο, θα μπορείτε και αυτό να το δείτε. Θα μπορείτε επίσης να δείτε ποια είναι η άποψη της ΕΟΚΕ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας σήμερα. Να περάσουμε τώρα σε πάνω από μία ώρα ψηφοφορία, γιατί έχουμε πάρα πολλά ε, έγγραφα να ψηφίσουμε. Ο εισηγητής είναι και πάλι ασχολημένος. I just check. So are you happy with Are you happy with that um? Συμφωνείτε με αυτά που είπα? Ωραία. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Θα χρησιμοποιήσουμε και τις ηλεκτρονικές μας κάρτες. Ελπίζω να τις έχετε όλοι. Πρώτη μας ψηφοφορία. Γνωμοδότηση της Evelyn Gebhardt. Εκβιομηχάνηση της Ευρώπης για την προγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας. Θέλετε να πάρετε το λόγο πριν από την ψηφοφορία, κυρία Gebhardt. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους μου, σκιώδεις συγητές. Εξεπλάγει λίγο. Ήταν πολλές, πάρα πολύ καλές και πάρα πολύ θετικές οι τροπολογίες ε, προς τη δική μου κατεύθυνση και θεώρησα ότι είχε νόημα να τις συνοψίσω. Γι' αυτό έκανα τις λεγόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες. Και τώρα ξαφνικά οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκό Κόμματος, ε, οι φιλελεύθεροι ε, και άλλη μία ομάδα θεώρησαν ότι αν δεν θέλουμε τις συμβιβαστικέ θα ψηφίσουμε τις αρχικές τροπολογίες. Και ξαφνικά ακούω ότι το ΕΛΚ θέλει να φέρει και προφορικές τροπολογίες. Ε, όχι, αυτό το παρατραβάει έχω συνεννοηθεί με τις τρεις πολιτικές ομάδες. Είπαμε να ψηφίσουμε τις τροπολογίες όπως έχουν κατατεθεί αν δεν θέλετε συμβιβαστικές. Πάντως τώρα προφορικές τροπολογίες δεν πρόκειται να δεχθώ. Θα έπρεπε να τα είχαμε συζητήσει αυτά στα πλαίσια ε, της εκπόνησης συμβιβαστικών τροπολογιών για να τα λύσουμε, αλλά έτσι δεν γινόνται αυτά τα πράγματα, παρακαλώ πολύ. Okay, well, thank you. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καταλάβαμε σαφής η θέση σας. Ε, δεν θα δώσω τη δυνατότητα προφορικών τροπολογιών, γιατί όπως ξέρετε μόνο με τη συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων μπορούν να υποβληθούν και δεν θα ήθελα να αρχίσουμε συζήτηση γι' αυτό και θα χρειαστούμε όλο το πρωινό. Ας πάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Τέλος πάντων αυτό είναι ένα μάθημα για την επόμενη φορά. Τροπολογία 2. Έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία, παράγρα, ε, συγγνώμη, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, απο, Ποιες εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για να δούμε κατά πόσο δουλεύει το σύστημα για το δεύτερο τμήμα. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 13-20. Καταπίπτει η τροπολογία 1. Ψηφίζουμε την τροπολογία 3. Προσθήκη μία λέξη Την τροπολογία 3 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 5 υπέρ. Να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 5. Έναξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20-14. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 11. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Είναι επίση μία προσθήκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13. Έναρξη ψηφοφορία ηλεκτρονικό για τη 13. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρα... Επειδή καταψηφίσαμε τη 13, Τώρα πάμε στην ε, τροπολογία 15 χωρίς την προφορική τροπολογία. Λοιπόν, υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Κατά τμήματα ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφέστατα. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται επίσης. Τροπολογία 12 ως προσθήκη στη 14. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 16 Όμπερμαϊερ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά απορρίπτεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 20 προσθήκη στη 17 υπέρ κατά απορρίπτεται 8 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 21 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος. τη 21. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 18-17. Τροπολογή 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24. Ως προσθήκη υπέρ κατά, εγκρίνεται. 22, επίσης προσθήκη, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 23, ε, ως προσθήκη, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 27, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 26, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 31, υπέρ, κατά εγκρίνεται 28. 28 χωρίς την ε, προφορική τροπολογία. 28 χωρίς την ε, προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 34, 33 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 34 υπέρ. Καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς την τροπολογία 34. Έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, απορρίπτεται. 16-19. 37. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τώρα τα 37 υπέρ. Καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικός την 37. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας απορρίπτεται 16-18. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Σε αυτή την περίπτωση 38 καταπίπτει. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στη 36 μου λέτε. Ωραία. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 20-15. 36 εγκρίθηκε, 38 και 41 καταπίπτουν άρα. 39 καταπίπτει επίσης. Όμως η 35 να ψηφίσουμε 35 ως προσθήκη. Κυρία Γκέπχαρτ, συμφωνείτε. Ωραία. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη 35. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. 40. Ως προσθήκη. Το στά, κυρία Γκέπχαρτ. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Εντάξει, ηλεκτρονικός να ψηφίσουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά εγκρίνεται. 48 έχει αποσυρθεί. 47 υπέρ κατά εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά εγκρίνεται. 51 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. 40 49. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης. Ηλεκτρονικώς θα ψηφίσουμε για τα πρακτικά. Έναρξη ψηφοφορίας για το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης. Πέρας. Εγκρίνεται. 21-3. 11 αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Say anything? Yes. Ε, κυρία Γκέπχαρτ. Θέλω να πω κάτι. Ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία. Εγώ σύστησα στην ομάδα μου αποχή. Όχι γιατί χάλασε η έκθεση ξαφνικά, αλλά γιατί ένα μεγάλο τμήμα εκείνων που ήταν απολύτως απαραίτητα για να υπάρχει μια συνολική θεώρηση της βιομηχανίας που είναι το εργατικό δίκαιο και τα κοινωνικά δικαιώματα. Βγήκαν από την έκθεση από την ε, συντηρητική και φιλελεύθερη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες δεν μπορούμε να τα δεχτούμε αυτά και ελπίζω να διορθωθούν στην καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή της Ουσίας. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος έτσι κι αλλιώς. Αυτό που πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε είναι η θέση μας αυτή που ψηφίσαμε να εκπροσωπηθεί και στην Επιτροπή Βιομηχανίας και είμαι βέβαιος ότι θα την εκπροσωπήσετε εξ ονόματός μας. Uh, European... Και τώρα ερχόμαστε στην έκθεση του κυρίου Γκαρσές Ραμόν. Θέλετε να πείτε τίποτα κύριε Σιγητά. Ε, μια νέα ατζέντα για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών. Περνούμε αμέσω λοιπόν στη ψηφοφορία. Θέλω να σας πω ότι Έχουμε βάλει πολλούς υποτίτλους για να βελτιωθεί το ευανάγνωστο της έκθεσης. Θα τα δείτε στην πορεία, ε, στον κατάλογο ψηφοφορία. Ε, ε, ψήφι υπέρ της προφορικής 1, κατά εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 91 ως προσθήκη υπέρ, κατά εγκρίνεται. 91 ως προσθήκη. Πέρας, εγκρίνεται, 28-6. Η τροπολογία 92, ψήφι πέ Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Η τροπολογία 90, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 85 καταπίπτει και οι υπόλοιπες. 93 ψήφι πέ Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 95 Τη κυρίας Καλιέτε σε τμήματα, τμήμα πρώτον, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 98, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 97 ως προσθήκη, υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 99 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 100 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 103 προ τίκη. υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά εγκρίνεται. 106 ως προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται. 108 υπέρ. Αυτό θα χρειαστεί ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. 108 ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. 17-17. 107. Τώρα μπορούμε να την ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Δεν είναι πολύ σαφές. Μήπως να σηκώνατε κανένα χέρι. Είτε λοιπόν ηλεκτρονικός. Πέρας. Εγκρίνεται 22 υπέρ 12 κατά. 109 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 110 υπέρ. Υπέρ. κατά. 111 υπέρ. 112 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Η συμβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται η συμβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι χρειάζεται να το ελέγξουμε αυτό. Uh, Απορρίπτεται. 17 υπέρ 18 κατά. 128. Αυτή ψηφίσαμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ και πάλι θέλει έλεγχο 133 παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση Votes closed. Uh, that's Πέρασε. 131 κατά έτσι δεν είναι, 131 καταπίπτει. Μπορούμε να ψηφίσουμε ως προσθήκη όμως την 132. Ψήφι υπέ, προσθήκη. Κατά, εγκρίνεται. 130 επίσης ως προσθήκη. Α, όχι, όχι, έχει καταπέσει, διορθώνει ο πρόεδρος. 135, ψήφι υπέ. Κατά, εγκρίνεται. 134 υπέ. Κατά, εγκρίνεται. 136 έχει αποσυρθεί. Η προφορική 2 υπότιτλος ψηφίπε κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 Είπε. κατά εγκρίνεται. 142 Είπε. κατά εγκρίνεται 141 Είπε. κατά εγκρίνεται 143 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται Προφορική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται σαφέστατα. Και θα περάσουμε τώρα στην 150 της κυρίας Γκέπχαρτ, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άλλος υπότιτλος υπέρ, κατά, δεν είναι σαφές. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ελέγχουμε την προφορική τροπολογία παριθμών 4. Αρχίζει ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε, πάμε στην 154 ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 πε. Κατά εγκρίνεται. 153 πίπτη, 156 επίσης. 158 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 157. Αυτό τι είναι τώρα εδώ προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προφορική 5. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι για τον υπότιτλο τι λέει καταναλωτές. Απορρίπτεται με ισοψηφία 17-17. Ε, συμβαστική 5 υπέρ, κατά. Σαφέστατα εγκρίνεται. Και τώρα έρχομαι στον υπότιτλο 6. Δικαιώματα επιβατών. Αρχής ηλεκτρονική ψηφοφορία. Καλά, δεν ήξερα ότι και οι υπότιτλοι είναι τόσο επίμαχοι. Πέρας. Απορρίπτεται με δύο ψήφους ο υπότιτλος. Ζητώ συγγνώμη προς τον εισηγητή. Δεν βρίσκουν εύνοια υπότιτλοι σας σήμερα, είπε. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7, είπε κατά άποχες εγκρίνεται και πάμε στην 179 στην αρχή της σελίδας πάνω πάνω στη 12 υπέ της 179 του κυρίου Πουπάκη κατά απορρίπτεται προφορική 7 για υπότιτλο υπέ αυτή θα περάσει μάλλον η επικεφαλίδα. Εντάξει, εγκρίνεται. 182. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 181 καταπίπτει. 183 και 84 μαζί υπέρ. Ταυτίζονται. Κατά. Εγκρίνονται. 187 και 186 και 185 καταπίπτουν. 188 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 8 υπέρ κατά σαφώς εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβαστική 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και τώρα η 197 198 197-198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 200 ψήφι υπέρ κατά εγκρίνεται. Προφορική 9 υπέρ. Α, αρχίζει η ψηφοφορία. Άλλος ε, ε, αμφιλεγόμενος υπότιτλος. Αϊφόρος κατανάλωση. Πέρας. 16 υπέρ 19 κατά. Πάλι έχασε και αυτό η φέλιδα. <laughs> Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε σαφείς υποτίθεση, τελικά. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 202 ως προσθήκη στη συμβαστική 10 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 208 έχει αποσυρθεί και πάμε να σας πω αμέσως ε, στη 209 ψήφι υπέρ γιατί και 208 έχει αποσυρθεί είπαμε ε, υπέρ της 209 ε, κατά εδώ χρειάζεται έλεγχος ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 209 παρακαλώ αρχίζει η ψηφοφορία Απορρίπτεται. 2.11. Ροσπόρ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 210 κατά πίπτη. 2.12. Υπέρ. Κατά. Α, δεν είναι σαφές καθόλου όμως. Ψηφίζουμε την 212, ε, παρακαλώ. The vote's closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 17-18. Καθυστερείτε πολύ στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ ψηφίστε πιο γρήγορα. 2-13. Η ψηφοφορία αρχίζει τώρα ηλεκτρονική. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Και τώρα η τελογική σκέψη. 23 τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά εγκρίνεται. 26, 24 πίπτων, 27 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 29 ως προσθήκη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 ως προσθήκη υπέρ, κατά εγκρίνεται. Η 31 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Η 38 έχει καλυφθεί από την 31, αλλά η 38 έχει και ένα δεύτερο τμήμα, αντίστοιχο που πρέπει να ψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 32 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 37 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 48 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 51. Μόνη της υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 49. Τι λέει εδώ, οριζόντια τροπολογία. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι σημαίνει οριζόντια τροπολογία. Α, καλύπτει διάφορα. Εντάξει. Ε, παρακαλώ ψηφίσουμε την οριζόντια τροπολογία της κυρίας Πίτη Κάινεν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται οριζόντια όμως. Η 50 αυτόματα εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 ψήφι Το πρώτο τμήμα, συγγνώμη. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Εγκρίνεται επίση. Και τώρα θα έρθουμε στη συμβαστική 14. Έτσι δεν είναι. Συμβαστική 14 ψήφι Κατά. Εγκρίνεται. Και η συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται επίσης. Η τροπολογία 68, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 69 και 71 μαζί, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 70 κατά πίπτη. Συμβιβαστική 17 ψήφι υπέρ, κατά εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά εγκρίνεται ή 78 της Επιτροπής Μεταφορών ως προσθήκη ψηφιπέ κατά εγκρίνεται 84 των μεταφορών υπέ κατά εγκρίνεται Η συμβιβαστική 19 υπέ κατά εγκρίνεται ή 79 υπέ. Νομίζω χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε την 79 παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται 20 υπέρ 14 ε, κατά η 80 του εισηγητή υπέρ υπέρ κατά νομίζω με την ίδια πλειοψηφία αλλά χρειάζεται έλεγχο ψηφίζουμε την 80 ηλεκτρονικός πέρας εγκρίνεται 21-13 Λοιπόν, τώρα είμαστε στι αιτιολογικές αναφορέ. Τροπολογία 1, ψήφι Κατά. Εγκρίνεται. 2. Ως προσθήκη. υπέ, Κατά. Α, όχι και πάλι χρειάζεται παλήθευση αυτό. Αρχίζει για τη 2. Του Jean-Pierre Οντί είναι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 3 υπέρ Κατά. Δεν είναι σαφέ. Το ΕΛΚ δεν ψηφίζει. Α, ψηφίζει τώρα. Η τρία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Η τέσσερα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η πέντε έχει αποσυρθεί. Και η έξι. Επτά υπέρ. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι την επτά. Πέρασε. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τις υπόλοιπες μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί 8, 9, 10 της Επιτροπής Μεταφορών. Ο συγητής τι λέει. Μπορούμε, ωραία. 8, 9, 10 τραν μαζί. Όχι. Γιατί όχι. 7 υπέρ, κατά. Την 7 την ψηφίσαμε. 8 λοιπόν. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά και αυτή εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά Υπέρ ξανά. Η τροπολογία 15 της κυρίας Ράπτη. Υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε τη 15 της κυρίας Ράπτη. Πέρας. Εγκρίθηκε 20-16. Η 16 έχει αποσυρθεί, τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 18 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά εγκρίνεται η 19 κατά πίπτη 20 υπέρ κατά νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά στην ελέγξουμε καλύτερα την 20 για καλό και για κακό απορρίπτεται 17 υπέρ 19 κατά. Η τροπολογία 21 αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικός για την 21. Πέρας. Με την ίδια πλειοψηφία, 17-19 απορρίπτεται. Ωραία. Το σύνολο της πρότασης γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικός αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Όχι. 36 ψηφίζεται με κάρτες, δεν ψηφίζεται. Πέρας. 34 υπέρ, 2 κατά, χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Γκαρσές Ραμόν. Πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Right, we now move on to my own report. Και τώρα ψηφίζουμε τη δική μου έκθεση γνωμοδότηση για την Επιτροπή Μεταφορών. Υπάρχουν διάφορες unblock ε, ψηφοφορίες, θα σας λέω κάθε φορά. Η πρώτη ψηφοφορία είναι μπλοκ για διάφορες τροπολογίες που θα αλλάξουν από αυτό από κανονισμό σε οδηγία. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκαέξι μέχρι 100 Ποιοι είναι υπέρ αυτής της αλλαγής, κατά. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Κύριε Αμάντερ. Ο κύριος Φαπ. Πρόεδρε, μπορείτε να πείτε ποιες είναι οι επιπτώσεις της ψηφοφορίας στο να γίνει ο κανονισμός οδηγία δεν θα έχει καμία αρνητική επίπτωση για την ενιαία αγορά. Μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε αυτό παρακαλώ. Συμφωνώ, ναι. Πάμε στην 39 του κυρίου Βαντεκάμπα. Υπέρκατα εγκρίνεται. Τώρα έχουμε ένα άλλο, μια άλλη unblock ψηφοφορία από διάφορους ε, ε, συναδέλφους με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν τα μοτοσακά από το πεδίο εφαρμογή 41, 42, 47, 48 και 57. Είναι σημαντική η αυτή η ψηφοφορία. Είναι, όπως σας είπα, unblock. Ώστε να βγουν τα μοτοσακά από το πεδίο εφαρμογής. Ψηφίζουμε. 42, 43, 44, 47, 48, 50 και 56, 57. Όλες αυτές μαζί. Εντάξει, καταλάβατε όλοι. Ξέρω ποιοι είναι κατά. Η κυρία Βέσφαλ είναι κατά, μου το είπε και χτες. Οπότε, Είπαμε, είναι για να φύγουν τα μοτοσακά από το πεδίο της οδηγίας. Ψηφίσατε, μοτοσυκλέτες. Η 58 καταπίπτει, γιατί εγκρίθηκαν όλες αυτές. Μετά έχουμε άλλη μια σειρά. Τροπολογίες 3, 4, 5, 6 και 7 που αλλάζουν τον ορισμό του αυτοκινήτου Αντίκα. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτοκίνητα αντίκε. Είναι το πακέτο εδώ. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται, εγκρίνονται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 51 καταπίπτει και πάμε στην 52 Βέστφαλο υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 54 έχει αποσυρθεί συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 ε, 5 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην τροπολογία 61 Βέστιφαλ. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Και μετά έχουμε την τροπολογία 63 ως προφορική τροπολογία που είναι από, την, από τον κύριο Μάντερς. Η προφορική υπέρ κατά εγκρίνεται. Εγκρίναμε την 63 λοιπόν με την προφορική μάλλον είναι η 63 της κυρίας Βέσφαλ με προφορική τροπολογία, 64 καταπίπτει και άρα πρέπει... Όχι, πρέπει να ψηφίσουμε και για την 64. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Καταπίπτει. Τροπολογία 11 υπέρ κατά εγκρίνεται, 70 υπέρ κατά εγκρίνεται, 73 μάντερς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην 85, Βαντεκάμπ, υπέρ, κατά, ε, εγκρίνεται, τροπολογία 13, τεχνική προσαρμογή λέει εδώ θα γίνει. Τροπολογία 14, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, γιατί 13 δεν χρειάζεται Όχι, πρέπει να ψηφίσουμε για τη 13. 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τις επόμενες μπορούμε να τις ε, δούμε unblock, να τι ψηφίσουμε unblock, γιατί αφορούν όλες τεχνικές βελτιώσεις. Είστε Ωραία, έχουμε δηλαδή τις τροπολογίες του δεύτερου παρατήματος 15, 101 μέχρι και 109. Υπερκατά εγκρίνονται. Πάω τώρα στην τροπολογία 18 υπέρ κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 22 έχει καταπέσει 23 υπέρ κατά εγκρίνεται 24 υπέρ κατά εγκρίνεται 25 υπέρ κατά εγκρίνεται 26 έχει αποσυρθεί 27 υπέρ κατά εγκρίνεται 28 έχει αποσυρθεί τροπολογία 1 υπέρ κατά εγκρίνεται 29 έχει αποσυρθεί 30 έχει καταπέσει γιατί η 10 εγκρίθηκε ή όχι θα το δούμε άμα χρειαστεί λοιπόν ε, ε, η 2 υπέρ κατά εγκρίνεται 31 έχει καταπέσει 35 υπέρ κατά εγκρίνεται Λοιπόν, ψηφίζουμε για τελική ψηφοφορία για τη γνωμοδότησή μου. Ψηφίζουμε λοιπόν και σας καλώ να την υπερψηφίσετε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ, 7 κατά. Λοιπόν, Λυπούμε που δεν έψα τον κύριο Μάντρας να υποστηρίξει τη γνωμοδότησή μου, αλλά θα την υπερασπιστώ πέναντι στην Επιτροπή Μεταφορών. Σας ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν. Περνάμε τώρα στην οδηγία, στην αναδιατύπωση της οδηγίας για την διαμεσολάβηση των, ε, στις ασφαλίσεις. Εδώ είναι περίπλοκη η ψηφοφορία. Να προσέξουμε λοιπόν πολύ. Υπάρχουν και συμβιβαστικέ. Κυρία Στάιλερ, θέλετε να πείτε κάτι πριν να ψηφίσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με την 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 38. Τροπολογία 38. Σμιτ την έχει αποσύρει. Είμαστε τώρα στην τροπολογία 39. Καράς. Υπέρ κατά Τροπολογία 39. Καράς. Τέλος της πληροφορίας Απορρίπτεται. 40 χάρας υπέρ, κατά, ε, εγκρίνεται, με συγχωρείτε. Συμβαστική α υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 43 υπέρ, 43 υπέρ, κατά, Δεν βλέπω να σηκώνονται χέρια βασικά. Σας παρακαλώ λοιπόν λίγο να γυμναστείτε. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται λοιπόν. 44 υπέρ κατά απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογική. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έξι το εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. Έλεγχος. Τροπολογία έξι του εισηγητή. Απορρίπτω δεν Όχι, ε, καλά κάνατε και ζητήσατε έλεγχο. Τροπολογία 48, Σμιτ και Χατζημαρκάκης. «48 ψηφίζουμε τώρα. Τροπολογία 48. Τέλος της ψηφοφορίας. Ε, γκρίνεται. 49. Υπέρ. 49. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε για τη 49. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. Συμβαστική σε. Η συμβαστική καταπίπτει λοιπόν γιατί εγκρίθηκε η 49. Πάμε στην 51. 51, τροπολογία 51. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 του εισηγητή. τη εισηγητρίας. Με συγχωρείτε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17-17. Δύο δεν ψηφίζουν. Αν ψηφίσετε θα επηρεάσετε το αποτέλεσμα. 52 υπέρ κατά εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στη 56. Υπέρ. Πρέπει να ξεκινήσουμε ψηφοφορία τώρα γι' αυτό. 56. Τι ηλεκτρονικό έλεγχο εννοώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 57. Ψηφίζουμε για την 57. Απορρίπτεται με μία ψήφο. 18-17. Έχει διαγραφεί από τον κύριο Σμίτ υπέρ κατά εγκρίνεται. Μάλλον καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. γιατί υπάρχουν συνέπειες εδώ. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Εγκρίνεται, οπότε όλα τα άλλα καταπίπτουν στο άρθρο 4 και πάμε στην 62. So we are now on to Amendment 62. Those Τροπολογία 62 υπέρ κατά εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ υπέρ κατά απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά εγκρίνεται. 69 και 70 υπέρ κατά εγκρίνονται. 71 και 72 υπέρ κατά εγκρίνονται. 73 και 74 υπέρ κατά εγκρίνονται. 75 και 76 και 77 υπέρ κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 12 καταπίπτει 13 τώρα. τι συγγήτριας υπέρ υπέρ πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά εδώ. 13 της εισηγήτριας. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Και τώρα πάμε στη συμβιβαστική Ή, e, ε. την ψηφίζουμε ε, μαζί με μια προφορική τροπολογία στο, ε, στην ατολική σκέψη. Λοιπόν, ε, ε, ψηφίζουμε... Μπερδεύτηκα, δεν πειράζει τώρα. Ακυρώνουμε την ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν της συμβιβαστικής ή ε, e? κατά εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 81, 82 και 83. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 14 καταπίπτει. Συμβαστική F υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογίες 85, 86 και 87. Να ψηφίσουμε αν μπλοκ για όλες τις διαγραφές. Μέχρι και την 99. Εντάξει. Unblock λοιπόν υπέρ, κατά. Ωραία, πέρασαν όλες. Και αυτή ξεμπερδέψαμε και με τη 13. Και έχουμε τώρα τη, την 100 και την 101 που καταπίπτουν και πάμε στη συμβαστική G. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβα... Ε, τροπολογία 15 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται. 106 του κυρίου Σμιτ υπέρ. 106 Σμιτ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. vote's closed. That's carried by two votes, 19 to 17. Τέλος ψηφοφορίας συγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά, 19-17. Συμβιβαστική H. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 108 ε, Σμιτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 109 και 110 υπέρ κατά εγκρίνονται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά υπέρ της συμβιβαστικής I Το έλεγχο πρότεινε αλλά δεν, την συμβαστική, αλλά τώρα δεν είναι τμήμα της, δεν, δεν στηρίζεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική I. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται, οπότε πάμε στην 114, 15 και 16. Υπέρ. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Καταπίπτει. Και πάμε στα 117 και 18. Υπέρ. Το άλλο δεν υπέρ κατά ε, εγκρίνεται σαφώς. 119 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 18 καταπίπτει. Τροπολογία 19 της εισηγητρίας υπέρ. Και εδώ θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 120, 121 και 22 από κοινού. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 120, 21, 22. Τέλος της ψηφοφορίας. 123 και 24. Ποιοι είναι υπέρ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αν μπορούσατε να συντομεύετε λίγο για να τελειώνουμε. Απορρίπτονται. Τροπολογία 20 της εισηγήτριας υπέρ. Λοιπόν, τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 20. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 19 προς 16. 125, 126, 127. Ποιοι είναι κατά. Εγκρίνεται. 128 καταπίπτει, 129 καταπίπτει. Και πάμε στην 130, Σμιτ, υπέρ κατά, αποχε, ε, κατά εγκρίνεται. Συμβαστική K, υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 133, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 είναι συμβατή με την 133 της εισηγήτριας. Ε, ποιοι είναι υπέρ της 22. 22. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 134 Καράς Υπέρ Ηλεκτρονική ψηφοφορία Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά 135 υπέρ εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 23 της εισηγητρίας υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβιβαστική M υπέρ κατά εγκρίνεται. 142 και 43 υπέρ. Όχι. Αυτό να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε... Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με ισοψηφία. 144. Υπέρ. Και εδώ ας σπιβήσουμε ηλεκτρονικά. Εκατόν σαράντα πέντε υπέρ κατά απορρίπτεται 146, 47 και 48 υπέρ κατά εγκρίνονται συμβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται 24 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική ο υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 154 υπέρ 154. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 155. 155 δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται η 155 με μια ψήφο διαφορά. 156. Υπέρ κατά εγκρίνεται 157 υπέρ και αυτή εδώ η ψηφοφορία είναι τσίμα τσίμα ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά εγκρίνεται όχι, συγγνώμη, διορθώνει ο Πρόεδρος, απορρίπτεται. Συμβιβαστική π. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά εγκρίνεται. 160 καταπίπτει. 26 υπέρ ηλεκτρονική ψηφοφορία. 26 εγκρίνεται με μια ψήφο διαφορά. 160 καταπίπτει. 26 της εισηγήτριας. Α, τι κάναμε μόλις, ναι, σωστά. 162 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 165 και 66 υπέρ, εγκρίνονται. 67 υπέρ. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Εκατόν υπέρ κατά εγκρίνεται. Οπότε 169 καταπίπτει, 170 υπέρ. Και πάλι εδώ είναι τσίμα τσίμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 171. 171. Um, Ψηφίζουμε για την 171. but that's carried. 172. Those in favor. 172 υπέρ. Κατά εγκρίνεται ή 27 κατά πίπτη. 173, 74, 75 υπέρ. Και εδώ θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 173, 174, 175, the vote's open. Ψηφίζουμε. Απορρίπτονται. Τις επόμενες μπλοκ όχι. 176 ε, υπέρ, κατά εγκρίνεται. 177. 177. Ε, Ηλεκτρονικός έλεγχος. Uh, 177, Uh, Απορρίπτεται. 178. Ηλεκτρονικός, ε, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Same. But you can never tell. That's closed. Το ίδιο. Απορρίπτεται. 179. Πάλι ηλεκτρονικά. Να ελέγξω, ο και κανεί αλλάξει γνώμη εδώ μεταξύ. Απορρίπτεται. 180. 180. Votes open. Closed. Same. We could have done all these on blocks. 181. 181. Μπορεί ένας να αλλάξει γνώμη και να αλλάξει και το αποτέλεσμα. Για κάποια από όλες αυτές. Ορίστε, πάνω που το είπα. Μία ψήφο διαφορά και πέρασε. Καλά που χρησιμοποίησαμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. 182 τελευταία από αυτές. Για να δούμε θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται τι; Ωραία λοιπόν. Πάμε τώρα στα εκτιμώντας. Λοιπόν, το εκτιμώντας 28 έχει ήδη εγκριθεί γιατί εγκρίναμε τη συμβαστική νωρίτερα. Πάμε στην συμβαστική Q. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 30 καράς Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Του εισηγητή. Τη εισηγήτρια, με συγχωρείτε. Τέλος. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο. 31 κάρας ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Τροπολογία 2 της ηγητρίας. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ρο υπέρ κατά εγκρίνεται επόμενες τρεις unblock. Αρχίζουμε την ψηφοφορία για τα επόμενα 33, 34, 35 και 36 λοιπόν μαζί. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας και απορρίφθηκαν. 17 υπέρ, 17 κατά. Και τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο της γνωμοδότησης. Εγκρίνεται 34 ψήφοι πέρα και μία κατά. Κυρία Στάιλερ, σαφής η εντολή μας να υπερασπιστείτε τη θέση μας. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι. Ωραία. Τελευταία ψηφοφορία λοιπόν για σήμερα. Είναι η έκθεση του κυρίου Παντσέρη για βασικές πληροφορίες, έγγραφα με βασικές πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά προϊόντα. Ο κ. Παντζέρη δεν είναι εδώ. Περνάμε λοιπόν απευθεία στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται 5 υπέρ κατά απορρίπτεται 45 υπέρ κατά εγκρίνεται 46 υπέρ κατά εγκρίνεται 6 του εισηγητή υπέρ κατά απορρίπτεται 47 υπέρ κατά απορρίπτεται 6 υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 49. Συμβατή με την 8. Υπέρ. Είναι και η προφορική τροπολογία βεβαίως. Από την ΚΟΕ. Υπέρ κατά. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικό ωραία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Έτσι για να ξυπνάτε. Για τη 49. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική A. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Πρέπει να πάω προς τα πίσω. Επειδή απορρίφθηκε η τροπολογία με την προφορική τροπολογία, τώρα πρέπει να ψηφίσουμε αυτήν ε, που δεν έχει την προφορική τροπολογία, να δούμε αν θα περάσει αυτή. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική A. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική B. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 61 κατά πίπτη. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 65 ρούλε υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 12. Το εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 66. Χάντελ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 68 το συμβατεί με τη 13 υπέρ κατά εγκρίνεται 69 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική E υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική F υπέρ κατά εγκρίνεται πάμε λοιπόν στην τροπολογία 76 ρέπο συμβατή υπέρ Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 76. περασε εγκρινεται Εγκρίνεται. 22-13. 77. Υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Νομίζω ότι καλύτερα να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικό στην 77. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να είμαστε σίγουροι. Εγκρίνεται 21-13. 78 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 84 Χέντελ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 85 Πιετικά είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 86 Χάντελ υπέρ Κατά. Απολύπτεται. Άρα, 87 Σμιτ υπέρ. Υπέρ, κατά. Καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Την 87 άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 19, 14, 16. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά εγκρίνεται. 18 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 92 σμίτη έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 92. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική J υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική K υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. L υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 102 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 104. Μπουσόι, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 22 του εισηγητή, υπέρ, κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά τσίμα τσίμα. Να ξαναψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικό στην 22. Πέρας εγκρίνεται. 105. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. 106. Λοιπόν, εγώ έχω μπερδευτεί τώρα εδώ. Έχει προφορική τροπολογία από την Άλντε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 107-108 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική M υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Έναρξη ψηφοφορία για την 111. Δεν έβλεπα καλά. Πέρας. Εγκρίνεται. 112. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24 του εισηγητή. Υπέρ. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικό. Στην 24 νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρας. Εγκρίνεται 21-14. 113 μάντερς. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική N. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική O. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφέστατα. Λοιπόν. Τώρα που πάμε. Στην 139. Ωραία. Σμιτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Υπέρ κατά εγκρίνεται 144 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 145 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 146 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 147 υπέρ. Κατά Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Κύριε Σμιτ, τα καταφέρατε. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές αναφορές. 26, Γιατί κάνει υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 27, Χάντελ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 28. Του εισηγητή υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 29 Χάντελ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 30 με την προφορική τροπολογία. Χάντελ, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 30 χωρίς την προφορική τροπολογία, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 31, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 32, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 33, ως προστίκη, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 34, μπουζόι, υπέρ κατά εγκρίνεται 35 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική π υπέρ κατά εγκρίνεται 39 υπέρ κατά εγκρίνεται 40 υπέρ κατά απορρίπτεται 41 υπέρ κατά εγκρίνεται 42 υπέρ κατά, απορρίπτεται και 43 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικός, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. right. Εγκρίνεται 34 ένα. Συγχαρητήρια κύριε Παντσέρη και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ολοκληρώνονται εδώ οι σημερινέ ψηφοφορίε. Σα ευχαριστώ πολύ και σα ευχαριστώ για την έντονη προσοχή που δείξατε όλη αυτή την ώρα. Έχουμε μόνο πέντε λεπτά καθυστέρηση. Η κυρία Κόρατσα Μπίλτ την επόμενη σημερινή σε διάταξη. Θα αφήσουμε ένα-δύο λεπτά να φύγουν όσοι δεν θέλουν να παραμείνουν πριν παρακαλέσω την κυρία Κορατσαμπίλτη να λάβει το λόγο.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 την επόμενη συζήτησή μας, που είναι η έκθεση πρωτοβουλίας ε, της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ. Είχε γίνει και μια πολύ επιτυχής ακρόαση για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών, περιγραφή της κατάστασης και επόμενα βήματα. Έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης να εξετάσουμε το οποίο θα μας το παρουσιάσει η εισηγήτρια. Έχουμε σκιώδεις εισηγητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Λόκεγκαρτ είναι εδώ, η κυρία Ράπτη όμως δεν είναι εδώ, δεν ξέρω ποιος θα την αντικαταστήσει η κυρία Γκέπχαρτ ενδεχομένω. Θα την καταστήσετε την κυρία Ράπτη. Μάλιστα. Ωραία. Ρούλε, η κυρία Ρούλε και εγώ. Η Κλέρ είναι εδώ με τους συνεργάτες της ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα της δώσω το λόγο ε, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησής μας. Ε, Άννα Μαρία, σου δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσεις την έκθεσή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι εδώ ε, μια ομάδα επισκεπτών από την Καλσκούγκα. Θα ήθελα να τους, από τη Σουηδία, ε, από τον... Ε, Εμείς είμαστε ε, ο οίκος των Ευρωπαίων πολιτών, οπότε καλώς ήρθατε. Το θέμα λοιπόν ε, αφορά ε, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 70% του ΑΕΠ και της απασχόλησης προέρχεται από την αγορά υπηρεσιών, που είναι ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας. Θα μπορούσαμε 330 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,6% του ΑΕΠ να έχουμε σε 5 με 10 χρόνια αν αναπτυσσόταν πλήρως το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς ε, ή υπηρεσιών. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν η Προεδρία ε, ή κάποιο κράτο μέλος ε, είναι παρόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε, μια, έχουμε ιστορικά ποσοστά ανεργίας πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για πολύ, λίγη, για πολύ λιτότητα και λίγη ανάπτυξη. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι κυβερνήσεις θεωρούν ότι οι εθνικές πολιτικές είναι επαρκείς για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη ή αν ο αυτός είναι ο τομέας στον οποίο θα μπορούσαμε ε, χωρίς ε, δαπάνη, δαπάνες ε, των χρημάτων των φορολογουμένων να αναπτύξουμε τον τομέα των υπηρεσιών. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν. Έχουμε μία ε, οδηγία υπηρεσιών που εγκρίναμε το 2006 και θα ήθελα να χαιρετήσω το ρόλο της κυρίας Γκέπχαρτ, ε, της κυρίας Χάντζλικ ε, και του δικό σας κύριε Πρόεδρε και άλλων συναδέλφων βεβαίως με ιδιαίτερη αφοσίωση από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή. Έχει μεταγραφεί, αλλά δεν ε, επιβάλλεται η εφαρμογή της πλήρως. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν ε, στα, τα κράτη-μέλη πώς εξηγείτε στους πολίτες σας ότι τους στερείτε θέσεις απασχόλησης που δεν ε, στοιχίζουν δημόσια χρήματα και θα ήθελα να είστε πιο υπόλογοι και πιο διαφανείς σε αυτή τη διαδικασία σε σχέση με εμά τι ακριβώς δεν εφαρμόζεται, να είμαστε συγκεκριμένοι. Αν αγοράζει κανείς ένα πακέτο ταξιδιωτικό από ένα κράτος μέλος, ε, μπορεί να τύχει κανείς διακριτικής μεταχείρισης λόγω του διαβατηρίου του. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καταναλωτών που είναι σήμερα εδώ για να μας πούν ότι επιλύθηκε η υπόθεση των Αυστριακών καταναλωτών που τους ζητήθηκε να πληρώσουν πολύ περισσότερα για ακριβώς την ίδια κρουασιέρα με αυτή που έκαναν Γερμανοί ε, ταξιδιώτες. Ε, άρθρο 22, ε, διάκριση με βάση την εθνικότητα και χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάση με τα κράτη-μέλη για να δώσει στους καταναλωτές της Ευρώπης να απολαύσουν πλήρως ε, την αγορά των υπηρεσιών χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις. Και οι εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ε, μια αγορά 500 ε, εκατομμυρίων ατόμων αν, ας πούμε, ένας αρχιτέκτονας θέλει να έχει επαγγελματική δραστηριότητα σε μια άλλη χώρα, πρέπει να δείξει ότι 51% ε, της εταιρείας του ανήκει σε ιδιώτες ή αλλιώς πρέπει να αλλάξει τη νομική μορφή της εταιρείας. Ή ας πούμε μια, ασφαλιστική, μια εταιρεία που έχει ήδη μια ασφάλεια και θα μπορούσε να υποχρεωθεί να πάρει μια ακόμη ασφάλεια, δηλαδή διπλό κόστος για να μπορέσει να εγκατασταθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος. Και χαίρομαι ε, για τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το θέμα αυτό. Οι ασφάλειες πρέπει διασυνοριακά να αναγνωρίζονται. Θα μπορούσα να συνεχίσω με πάμπολα παραδείγματα αλλά η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τα ανέφερε. Τι κάνουμε. Υπάρχουν οι κανόνες. Η δουλειά μας είναι να ε, εξασφαλίσουμε ότι σωστά και με κατάλληλο τρόπο ε, εφαρμόζονται. Το πρόβλημα είναι στο τμήμα της αγοράς της οδηγίας υπηρεσιών όπου, υπάρχουν τα, όπου τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο ερμηνείας. Πολλές φορές, πολύ συχνά, ο λόγος του δημοσίου, ο λόγος του δημοσίου συμφέροντος ε, ερμηνεύεται με κάποιο τρόπο που δημιουργεί προσκόμματα. Ε, ζητώ λοιπόν στην έκθεσή μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει να διευκρινίσουμε, να καθοδηγήσουμε τα κράτη-μέλη για ε, το πώς θα εφαρμόσουν τον έλεγχο αναλογικότητας. Επίσης, η ε, ελεγχη οικονομικων οικονομικών αναγκών, δηλαδή ζητούν ε, κάποια κράτη-μέλη από άλλες χώρες να εξηγήσουν κατά πόσο υπάρχει προστιθέμενη αξία. Όλα αυτά τα πράγματα ε, στερούν θέσεις απασχόλησης από τους πολίτες μας. Στη δουλειά μας είναι σημαντικό να λέμε ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε δύο μέτρα και σταθμά. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν κοινή ευθύνη για το άνοιγμα των αγορών τους. Έχουμε επίσης από το 2006 μια νέα κατάσταση για να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά υπηρεσιών το να ενισχύσουμε την αγορά υπηρεσιών την εσωτερική είναι πολύ επικερδές ε, και για τη βιομηχανία. Ε, γιατί μπορούμε, έχουμε ας πούμε τις ε, κινητές υπηρεσίες, ψηφιακές υπηρεσίες, ε, συχνά ε, πολλούμε αγορά, υπηρεσίες και προϊόντα μαζί. Έχει πραγματικά εξελιχθεί τεχνολογία και μπορεί να αυξήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να απολαύσουν την εσωτερική αγορά οι πολίτες σε διασυνοριακό επίπεδο. Εναρμοσιμένη προσέγγιση και εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό με εναρμονισμένο τρόπο, Προσπαθούμε με εθνική νομοθεσία, τοπική νομοθεσία, ε, να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ιδάλλως, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση. Καλύτερη χρήση δηλαδή ε, του ε, συστήματος ενημέρωσης για την εσωτερική αγορά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το Solvit, που είναι ένας πολύ καλός μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Πρέπει να αναπτύξουμε τα σημεία επαφής δεύτερης γενεάς θα έπρεπε να είναι ένα πολύγλωσσο φιλικό προς το χρήστη, ε, φιλική προς το χρήστη δικτυακή πύλη για τους καταναλωτές και τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, τα καταστήσουν γνωστά διασυνοριακά. Θέλουμε να γίνει μια αξιολόγηση των ε, συγκριτικών δικτών, των benchmarks. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους εμπειρογνώμονες από τη Σουηδία για το πώς θα μπορούσαν ε, τα single, point, ε, τα single contact points να αποτελέσουν ε, βασικό μοχλό. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς δύο μέτρα και σταθμά, είναι σημαντική ε, όταν μιλάμε για παραβίαση κανόνων. Πρέπει επίσης ε, να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, διάλογος μεταξύ τοπικών ε, εθνικών αρχών αλλά και μεταξύ κοινοβουλίου και κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση καλεί τα κρατημέλη να σε, σε, υψηλότερο, σε υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο, αλλά και καλούμε και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Έχω έρθει σε επαφή με την Ιρλανδική Προεδρία Θέλουμε λοιπόν να ζητήσουμε να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για η εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών όσο χρόνο και αν χρειαστεί αυτό και το λέω αυτό το είπε και ο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πρέπει να είναι τέλο πάντων ε, μια προτεραιότητα και στις, ε, στα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών. Θέλουμε έναν συγκεκριμένο χάρτη πορείας για την άρση των εμποδίων ε, στην προώθηση της απασχολησιμότητας στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα συγκεκριμένα. Έχουμε τι μελέτε ομοτήμων, τα peer reviews. Έχουμε τώρα, επειδή είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ε, συγκεκριμένες ε, ειδικέ αναχώρασης τάσης. Ε, είναι μια δουλειά μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να είναι ανοιχτά και διαφανή όλα αυτά που κάνουμε, να γνωρίζουμε ποια είναι τα κρατημέλη που δημιουργούν προβλήματα, ποιοι είναι οι περιορισμοί, ποια είναι τα εμπόδια. Ζητούμε λοιπόν περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη διαφάνεια ε, για τα ε, προσκόμματα που παραμένουν στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσω με πολύ χαρά και εσά και τους υπόλοιπους σκιώδης ηγητέ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την σαφή ε, έκθεση και τώρα θα καλέσω τους σκιώδες να συμβάλλουν ε, με αυτές τις εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας υπάρχει περιορισμός στον χώρο, ε, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλουν να προσθέσουν οι συνάδελφοι. Γκέμπχαρτ πρώτα, που είναι αντικαθιστά την σκιώδη εισηγήτρια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματο κυρίας Ράπτη. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να πάει στη Λισαβόνα. Ξέρετε, σήμερα η μεγάλη επέτειο στη Βορτογαλία. Ε, είναι εκεί για την επανάσταση των Γαριφάλων. Ε, ε αλλά χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να την εκπροσωπήσω. Με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ το θέμα. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ράπτη. Και ε, συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι αυτή η οδηγία είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την εσωτερική αγορά. Αλλά θέλει επίσης να θυμίσει ότι δεν είναι αυτός σκοπός. Και αν θέλετε να πω και δύο λόγια εξ ονόματος, όχι της κυρίας ράπτη, αλλά προσωπικά να πω, κυρία Κοράτσα, συνέχεια μας πετάτε διάφορα νούμερα δεξιά και αριστερά εδώ και πάρα πολύ ψηλά. Μπορείτε να μας δίνετε και τις πηγές σας καμιά φορά. Γιατί ως εισηγήτρια εγώ ε, είχα πάρει πάρα πολλά αριθμητικά στοιχεία που δεν ήταν πάντα τεκμηριωμένα και στοιχειοθετημένα. Μιλώ για την οδηγία που είχα κάνει, θυμάστε, για τις υπηρεσίες. Δεν μου αρέσει αυτή η παπαγαλία διαφόρων ε, αριθμητικών στοιχείων που σας στέλνουν διάφοροι χωρίς να ξέρουμε πόθεν αυτά τα στοιχεία και τι αντιπροσωπούν. Η κυρία Ράπτη συμφωνεί ε, ότι χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας ε, για την παροχή υπηρεσιών και επίσης μετά από μία τετραετία, μετά το τέλος του χρονοδιαγράμματος που έπρεπε να έχει ακολουθηθεί, δεν έχει λήξει το θέμα. Πρέπει να γίνουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα. Μετά από τέσσερα χρόνια ελοπίσης δεν είναι ικατοποιητική η κατάσταση και ε, δεν ε, συμφωνούμε με τις καθυστερήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για μηδενική ανοχή και εσείς το ίδιο γενικά, όχι μόνο για το συγκεκριμένο. Ε, θα ήθελα να τονίσει επίσης η κυρία Ράπτη ότι ε, εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε ε, στην ε, σωστή υλοποίηση και στην ορθή εφαρμογή και όχι μία παρερμηνία ούτε διαστρέβλωση. Και αυτό που θέλουμε επίσης δεν είναι να τιμωρούμε τα κράτη-μέλη, αλλά να εξηγούμε όπου αυτό χρειάζεται και να βοηθούμε τα κράτη να εφαρμόζουν σωστά την οδηγία. Αυτό είναι πιο εύστοχο από οποιαδήποτε πειθαρχικά μέτρα και κυρώσει. Συμφωνεί ε, η κυρία Ράπτη μαζί σας ε, ότι αφορά την καλύτερη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς και βεβαίως μπορούμε να το συζητήσουμε όσο θέλετε και επίσης τις προτάσεις για τη διαφάνεια και την λογοδοσία. Accountability το λέει αυτό. Επίσης, συμφωνεί απολύθως μαζί σας η κυρία Ράπτη να διαδραματίζει ενεργό ρόλο και πρωταγωνιστικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά να δούμε και ποιο είναι ο ρόλος της προστασίας των καταναλωτών, να ενισχυθεί. Δεν μπορούμε να δεχτούμε διάκριση των καταναλωτών λόγω εθνικότητας, ηθαγένειας ή τόπου διαμονής. Το τονίσατε και εσείς αυτό. Και τα κράτη-μέλη και οι καταναλωτές αλλά και οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν ε, στην εφαρμογή. Υπάρχουν μερικά σημεία στα οποία όμως δεν μπορούμε να σας ακολουθήσουμε για να συμφωνήσουμε με την πρότασή σας κυρία Κοράτσα. Δηλαδή, εσείς θέλετε να πείτε ότι όλες οι εθνικές ρυθμίσεις είναι εμπόδια στην εφαρμογή της οδηγίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πει ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι εθνική ρύθμιση ε, ε, είναι απαγόρευση ή ανεπιθύμητη. Για να το ξανακοιτάξουμε αυτό παρακαλώ προσεκτικά. και να φροντίσουμε οι κανόνες που έχουμε θεσπίσει να εφαρμόζονται σωστά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταργηθούν ε, αμέσως ε, όλες οι εθνικές ρυθμίσεις και οι κανόνες. Ας πούμε, στο κοινωνικό και στο εργατικό δίκαιο και τα δικαιώματα. Και παρακαλώ την κυρία Κοράτσα να ξανακοιτάξει το άρθρο 20. Δεν έχει βγει η αρχή της χώρας προέλευσης. Είμαστε στη χώρα προορισμού. Δεν είναι μόνο το άρθρο 20, είναι και το άρθρο 1. Λοιπόν, θα πρέπει να ειδωθούν από κοινού αυτά. Γιατί εκεί ξεκαθαρίζεται ότι το εθνικό δίκαιο, ιδιαίτερα στην κοινωνική προστασία και τα εργατικά θέματα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Και αυτό. Για να υπάρχει μια κοινή βάση για συνεργασία που δεν θα πρέπει να λησπονούμε. Γι' αυτό η κυρία Ράπτη ακριβώς εδώ θα κάνει μια σειρά τροπολογιών και μόνο έτσι μπορεί να δεχτεί την έκθεσή σας. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί δυσανάλογοι, πραγματικά αυτοί θα πρέπει να καταργηθούν, συμφωνεί και η κυρία Ράπτη, αλλά με πολύ μεγάλη στάθμιση, ισορροπία και φρόνηση. Και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, θέλετε, να κάνετε πιο ε, ισορροπημένη την έκθεσή σας. Αυτή είναι η προσφορά για συνεργασία από την κυρία Ράπτη αλλά τα κοινωνικά δικαιώματα είναι σημαντικά, η προστασία των καταναλωτών, αυτά θέλουμε να τον νηστούν καλύτερα. Και μιλήσατε κι εσείς και για α, κάποιον στον οποίο θα πρέπει να απευθυνόμαστε και να ξέρουμε και ποιος θα είναι αυτός. Με ε, τροπολογίες θα τα επαναλάβουμε αυτά και εμείς γιατί νομίζουμε ότι είναι το κατεξοχήν σημαντικό θέμα. και πραγματικά εκεί χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία στα κράτη-μέλη. Γιατί αυτοί θα ανοίξουν τις πόρτες για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες που σε τελική ανάλυση δημιουργούν και τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Βλέπουμε λοιπόν πώς μπορούμε να ε, επιφέρουμε τη θέμενη αξία από τις εμπειρίες μας όσο προχωρούμε. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύτιμο το έργο σας, η έκθεσή σας. Κύριε Λόκεγκάρτ, ευχαριστώ πολύ. Ε, να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Κορατσαμπίλτ για την έκθεση. Είναι πάρα πολύ εύκολο για μένα να είμαι σκιώδης εισηγητής ε, σε αυτή την έκθεση, γιατί μου φαίνεται πολύ δύσκολο να διαφωνήσω μαζί σας τα κύρια σημεία. Οπότε θα ήθελα να πω ότι σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση. Υποστηρίζουμε πλήρως τη βασική ιδέα. Θα ήθελα επίσης σε τρία βασικά στοιχεία να τονίσω. Πρώτον, ότι, όπως είπε και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση στα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν τις προσπάθειές τους ε, για την εφαρμογή της οδηγία. Επίσης, υποστηρίζουμε την πολιτική μηδενικής ανοχής ε, για τις παραβάσεις ε, και την εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της νομοθεσία. Δεύτερον, συμφωνούμε απολύτω ότι είναι προβληματικό το γεγονός ε, ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος ε, χρησιμοποιούνται ως ε, αιτιολογία για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας. Τρίτον, μια σημαντική λεπτομέρεια σε σχέση με τη μη διάκριση για το άρθρο 22, το αναφέρατε κι εσείς. Συμφωνώ επί της αρχής ότι οι καταναλωτές δεν θα έπρεπε να την χάνουν διακριτικής μεταχείρισης ε, λόγω χώρας ε, διαμονής ή λόγω εθνικότητας. Όμως τα πράγματα είναι συχνά πιο περίπλοκα. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ότι οι επιχειρήσεις θα, μπο... θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν να πολλούν ε, στη Δανία και στη Σουηδία, για παράδειγμα, ή να μην θέλουν να πωλήσουν στη Γερμανία πρέπει να ακολουθήσουν τους καταναλωτικούς κανόνες της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Και το λέω αυτό και για τις μικρές και για τις μεσαίες επιχειρήσεις να γνωρίζουν το δίκαιο του καταναλωτή σε όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό το ζήτημα λοιπόν πρέπει να το αναφέρουμε στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης. Κάτι ακόμη. Συμφωνούμε απολύτως όπως είπα στα κύρια σημεία της έκθεσης ε, και αναμένω ένα γωνίο στενή συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Χάιντι. Πάρα πολύ σύντομα. Προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα γραπτό στα χέρια μας. Περιμένω να τελειώσει το σχέδιο έκθεση κυρία Κοράτσα και τότε θα συνεργαστούμε σίγουρα καλά. Κατά τα άλλα, ελπίζω να καταλαβαίνει και η ίδια ότι ως μικρή ομάδα δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να αφιερώνουμε σε γνωμοδοτήσεις. Δυστυχώς. Και πραγματικά θα την κάνω στον πόδι αυτή τη γνωμοδότηση. Σας το λέω από τώρα γιατί έχουμε τόσα πολλά νομοθετικά που δεν προκάνουμε σε μικρή πολιτική ομάδα να ασχολούμαστε με γνωμοδοτήσεις. Μα υπάρχει έκθεση, θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες νομίζω και θα φτάσει γρήγορα. Ε, μου λέγουν ότι έχει μεταφραστεί. Λοιπόν, να κάνω και εγώ μερικά σχόλια. Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που είπαν ότι είναι πολύ μεγάλη η δουλειά που έχει κάνει και έχει και περιορισμό σε σελίδες. Είναι έκθεση πρωτοβουλίας, ε, κυρία Κόρατσα. Ε, είναι πολλά τα σημεία που ε, θέλουμε να προσθέσουμε για να γίνει όσο ε, γίνεται πιο ολοκληρωμένη η έκθεση. Η δική μου βασική ανησυχία ποια είναι και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι σχετική έλλειψη προβολής των δυνατοτήτων που υπάρχουν σήμερα στην ενιαία αγορά σε ενδεχομένους επενδυτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και σε άλλες χώρες. Αλλά δεν προσαρμόζουν καν τα επιχειρηματικά του σχέδια, τα business plan που έχουν για να το πράττουν. Αυτό θα πρέπει να το πούμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται καλύτερο έλεγχο όλη αυτή η ιστορία. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν το προάγουν, δεν το προβάλλουν, δεν το διαφημίζουν. Έχουν κάνει επένδυση για να τα εφαρμόσουν όλα αυτά, για να τα υλοποιήσουν τα, τα ενιαία σημεία επαφής ή τη μεταφορά της οδηγίας και τη διαδικασία αξιολόγησης των νομοτήμων, αυτό το peer review. Πολύ μεγάλη επένδυση έχουν κάνει και σε συστήματα και σε προσωπικό για να φτάσουμε ως εδώ. Αλλά δεν το ε, κεφαλαιοποιούν αυτό το στοιχείο των επενδύσεων. Ας πούμε, δεν έχουν το όφελος που θα έπρεπε. Η οδηγία για τις υπηρεσίες ουσιαστικά τι έκανε. Μια σειρά από αλλαγές και μάλιστα ήταν καταλήτη ουσιαστικό για να κάνουν πολλέ λεπτομερεί αλλαγέ στα κρατημέλη στην εθνική του νομοθεσία. Τα λέει η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ε, παραμένουν αυθαίρετε απαιτήσει για ε, αδειοδότηση επιχειρήσεων που θέλουν να εγκατασταθούν στι χώρε. Για εγγραφή τους εμπορικά μητρώα, διάφοροι ε, λόγοι χρησιμοποιούνται ως πρόφαση δημοσίου δίθεν συμφέροντος για να προστατεύουν την εσωτερική αγορά των κρατών, την εγχώρια. Αυτά όλα θα πρέπει να ανήκουν στην ιστορία. Πολλές επιχειρήσεις προσπάθησαν να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα ε, και δεν ε, κατέστη δυνατόν τους. Βάζουν εμπόδια και ούτε το επιχειρούν ξανά γιατί θεωρούν ότι δεν αλλάζει τίποτα. Έχουν αλλάξει όμως τα πράγματα. Στην πραγματική οικονομία θα πρέπει να το δούμε. Πρέπει να, να, γίνει ορατό και εκεί. Αυτό που αναφέρει η κυρία Κοράτσα. Και ακριβώς εάν έρθουν οι υπηρεσίες αυτές από εταιρείε στα πλαίσια του νέου οικονομικού περιβάλλοντος, τότε θα υπάρξει πρόοδος. Κανονικά θα περίμενε κανείς να έχουν υλοποιηθεί όλα αυτά και κάποιες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και βλέπουν ε, δυσμενείς συνθήκες στη χώρα τους να θέλουν να ε, μεταφερθούν και σε άλλες χώρες. Αν δείτε τι γίνεται ε, με όρους Ανατολής Δύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Πολωνία αναπτύσσεται η οικονομία ε, και σε άλλες χώρες και ακολουθεί ένα μετασχηματισμό. Και πραγματικά χρειάζονται και ζητάνε αγωνίως ειδικού να του βοηθήσουν. Νέα πληροφοριακά συστήματα, ας πούμε, νέα συστήματα marketing. Χρειάζονται ειδικού. Προώθηση πολίσεων, ε, βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής, αναδιοργάνωση και μια σειρά άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο η αγορά των υπηρεσιών, αλλά και η πραγματική οικονομία που επωφελείται. Και μάλιστα είναι αμοιβαίως σε αυτή η σχέση. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε αυτή την προσπάθεια, να ενθαρρύνουν τις εταιρείε παροχής υπηρεσιών και αυτό δεν βοηθήσει μόνο τις υπηρεσίες αλλά το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και νομίζω ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νομοθετικό εγχείρημα και σχέδιο. Είναι μακρά η ιστορία της Επιτροπής μας σχετικά αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί για να μας απασχολεί, γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Αλλά ε, θα πρέπει να το μετασχηματίσουμε και να είναι ένα πραγματικό πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα ανάπτυξης σε επίπεδο και πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών. Με έχει καλέσει η Ιρλανδική Προεδρία να συμμετάσχω την άλλη εβδομάδα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας και θα υπάρξει συνεδρίαση για την περιφερειακή ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες και θα πρότεινα και με τη βοήθεια της κυρίας Κοράτσα να τα πούμε αυτά στους υπουργούς γιατί εκεί είναι η ευκαιρία αυτή και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Δεν πρέπει ίσως και σε άλλο κεφάλαιο να αναφέρουμε και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ε, των ενιαίων ε, για τη συνεργασία και την ε, επαφή με το κοινό και εκεί θα πρέπει να το αναβαθμίσουμε. Δεν θα πρέπει να αναβαθμίζουμε το υλικό, τους υπολογιστές ας πούμε να είναι δεύτερης γενιάς πιο σύγχρονης όταν δεν έχουμε πελάτες. Γιατί να αναβαθμίσω την υπηρεσία όταν δεν έχω σε ποιο να την πουλήσω. και τα στοιχεία για τη συγκριτική αξιολόγηση για την πραγματική χρήση όλων αυτών των δυνατοτήτων και την έκβαση τελικά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει για να δούμε πραγματικά ε, που θα οδηγήσουμε σε ένα νέο περιβάλλον. Um, on top of the other implementing data. So that's my... Um, και αυτή είναι η δική μου συνεισφορά. Λοιπόν, ποιο άλλο θέλει, ο κύριο Σφαπ, ο κύριο Λόκεργαρτ, ξανά, άλλο κανεί. Uh, so Mr. I'll invite Mr. Schwab and Mr. Lückegaard, and then I'm. I should have welcomed her very much earlier. Um, ε, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ο κύριος Σβάπ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι και καλωσορίζω την εισαγωγή της κυρίας Κοράτσα για το θέμα αυτό της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Είδαμε που θέλουμε να είναι το κέντρο βάρους και από κοινού και χωριστά. Και ελπίζω να καταλήξουμε και σε καλά αποτελέσματα. Να ξεκαθαρίσω από πλευράς του ΕΛΚ ότι και στις υπηρεσίες έχουμε μεγάλες δυνατότητες διασυνοριακής ανάπτυξης. Ήδη από σήμερα, είναι πολλά τα παραδείγματα, αλλά μπορώ να σας πω ότι ε, οι γερμανικές εταιρείες έχουν Ισπανούς μηχανικούς απορροφήσει και Ισπανούς αρχιτέκτονες ε, στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική. Ισπανούς που ήταν άνεργοι στην Ισπανία και ε, τελικά ε, εύκολα μπορούν να απασχοληθούν και κερδίζουν και καλά χρήματα. Δηλαδή και γι' αυτό μας βοηθούν αυτές οι ρυθμίσεις και τελικά είναι προς όφελος της παροχής υπηρεσιών και ε, είναι χρήσιμα και σκόπιμο. Η κυρία Κέπχαρτ μίλησε για τη διακυβέρνηση. Τι είναι αυτό το θέμα τώρα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα μη επίμαχα σημεία. Στη Γερμανία, ας πούμε, το θέμα της εκτίμησης των οικονομικών αναγκών έχει να κάνει ε, με τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες που πάνε και ανοίγουν ε, στην Ήπεθρο μεγάλα καταστήματα ε, λιανικής φθηνά, discount. Θα πρέπει να έρχονται σε επαφή όμως ε, με ε, την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι αρμόδια. Ε, δεν θα πρέπει να αποφασίζει για λόγους διακρίσεων, αλλά αν αποφασίσει ένας Δήμος ότι δεν θέλει να κάνει ένα τεράστιο κέντρο εμπορικό outlet δίπλα σε ένα αυτοκινητόδρομο, αυτό δεν είναι στρέβλωση του ανταγωνισμού, αυτό είναι χρήση γης και απόφαση για το πώς ε, θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει την επικράτειά του. Λοιπόν, θα πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλα τα προβλήματα εμπόδια και στρέβλωση του ανταγωνισμού. Θα πρέπει ε, να επικεντρωνόμαστε στα πραγματικά επίμαχα σημεία και στις πραγματικές δυσκολίες και εμπόδια και όχι στα φαινομενικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε να επανέλθετε, κύριε Λόκεγκάρτ. Ναι, να σας υποστηρίξω στις τελευταίες σας παρατηρήσεις. Νομίζω ότι πολύ σωστά τα είπατε. Αυτό που χρειαζόμαστε σε αυτή τη ε, συζήτηση είναι ενημερωμένα δεδομένα, νέα αριθμητικά στοιχεία που θα καταδεικνύουν τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορεί να βελτιωθεί. Μου φαίνεται δύσκολο να συμμετέχω σε συζητήσεις ακόμη και στη δική μου χώρα, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Χαίρομαι λοιπόν ε, που το εξετάζουμε ε, περισσότερο το θέμα, γιατί είναι κάτι το οποίο και εμένα μου απασχολεί πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Κλέρ, και μετά στην Αναμαρία Βαρατσαμπίλτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη του ε, στην ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ευχαριστώ πολύ την Ανά Μαρία ειδικότερα για την εξαιρετική τη ε, έκθεση, την οποία επικροτούμε. Είπατε κι εσείς ε, ότι είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός για τις επιχειρήσεις, για τους καταναλωτές, για τους ε, πολίτες μας, ε, αλλά και για λόγους κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα όταν είναι δύσκολη οικονομική συγκυρία. Χαιρετίζουμε το, την έκκληση προς τα κράτη-μέλη να δεσμευθούν πιο επικοδομητικά για πιο φιλόδοξη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών μέσω του διαλόγου με τα κράτη-μέλη και όταν χρειάζεται μέσω των επίσημων διαδικασιών αλλά και μέσω ε, επικοδομητικού διαλόγου και αναθεώρησης ομοτήμων ε, και, ε, να τα καταφέρουμε. Και όπως είπες και εσύ Μάλκολμ, πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε μια δυνατότητα πραγματική στις επιχειρήσεις ε, συμφωνώ με αυτά τα οποία τονίσατε και στην έκθεσή σας αλλά και στα σχόλια που ακούστηκαν σήμερα το πρωί. Για τα δεδομένα, γιατί αυτό αναφέρθηκε πολλές φορές, τα αριθμητικά στοιχεία της ε, έκθεσης της ε, κυρίας Μπίλτ βασίζονται στη μελέτη τη δική μας ε, από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς αλλά και με εμπειρογνώμονες ε, της ε, DG που είναι εμπειρογνώμονες στην οικονομετρία πώς θα καταφέρουμε μια πιο φιλόδοξη εφαρμογή της οδηγίας. Αν δει κανείς τα παραρτήματα της, κάθε χώρα, ε, ε, έκθεσης για την κάθε χώρα μπορεί να δει λεπτομέρειες για την κάθε χώρα. Αν θέλετε μπορώ να τις φέρω εγώ στο φως σαφέστερα ώστε να μπορείτε να τις δείτε. Τρία από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν. Πρώτον, για τους καταναλωτές. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει οι καταναλωτές ε, να μπορούν να νιώθουν τις συνέπειες εσωτερικής αγοράς. Ε, πολλές φορές ε, βλέπουμε καταγγελίες εμείς στη Γενική Διεύθυνση Μάρκτ όταν θέλουν να κάνουν μια ηλεκτρονική αγορά, για παράδειγμα, γιατί βρίσκουν ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση εναντίον τους. Ε, πρέπει και η Επιτροπή να μιλήσει στις επιχειρήσεις, να έρθει σε επαφή με τις επιχειρήσεις, αλλά και το Κοινοβούλιο πρέπει να το κάνει αυτό. Ε, Ξιότιμο συνάδελφό σας είπε ότι ε, δεν είναι αυτό η ουσία του προβλήματος. Ναι, αλλά εντάξει, μπορούμε να ε, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τις ε, επιχειρήσεις να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο. Όταν όμω ε, δεν βλέπουν τα ωφέλη της εσωτερική αγοράς, τότε πρέπει να έχουμε ένα διάλογο μαζί τους για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε. Το θέμα της αναλογικότητας ε, στη συνέχεια που αναφέρθηκε κάποιε φορέ. Η κυρία Γκέπχαρτ είπε, ε, είπε ότι η ρύθμιση δεν είναι αυτός σκοπός. συμφωνούμε με αυτό αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ψάξουμε και να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα που θα έπρεπε ο κανονισμός ε, να προστατεύει και αν είναι το κατάλληλο μέσο για να επιτευχθεί αυτό και θέλουμε να δούμε διάφορα ρυθμιστικά μοντέλα, όχι υποχρεωτικά γιατί θέλουμε να πούμε ότι κάποια είναι καλύτερα από άλλα, αλλά για να έχουμε μια καλύτερη επισκόπηση τη διαφορετική προσέγγιση, των διαφορετικών προσεγγίσεων, για να μπορέσουμε να κινηθούμε προ μια κατεύθυνση καλύτερη κατανόηση τη ε, αναλογικότητα. Ε, Όντω το είπατε αυτό και είναι σωστό ότι πρέπει να κάνουμε μια αναζήτηση για να το πετύχουμε. Τέλος, το θέμα της ε, πραγματικότητας ε, για τις ε, επιχειρήσεις. Ναι, όντως πρέπει να δαπανηθούν χρήματα, άρα τουλάχιστον να προωθήσουμε και αυτό που κάνουμε. Θεωρούμε ότι η δεύτερη γενεά του συστήματος πληροφόρησης είναι πολύ σημαντική, γιατί οι επιχειρήσεις θα πάνε σε ένα ενιαίο σημείο επαφής για να πάρουν τις πληροφορίες τους. Άρα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους. Και καταλαβαίνω ότι είπατε σε σχέση με τις προτεραιότητες, ίσως ο μήνας μια αγορά που θα έχουμε τώρα το φθινόπωρο θα είναι πολύ καλή ευκαιρία γιατί θα γίνουν πολλέ συζητήσει ε, και ε, στο διαδίκτυο αλλά και εκτό διαδικτύου να δούμε τι πρακτικά εργαλεία μπορούμε να αναπτύξουμε για τις μικρές επιχειρήσεις που όπως είπατε κι εσείς ε, πρέπει να έχουν συμμετοχή θέλουν να ξέρουν πώς μπορούν ας πούμε, να δραστηριοποιηθούν ε, ηλεκτρονικό στο διαδίκτυο και πρέπει να τις βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την έκθεσή σας. Νομίζουμε ότι πραγματικά λέτε τα πράγματα όπως έχουν και θα σας βοηθήσουμε όπως μπορούμε και εσάς και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ για την συνεχή υποστήριξή σου των προσπαθειών μας. Βεβαίω, είναι κοινέ οι προσπάθειές μας για να μπορέσει να προχωρήσει η αγορά υπηρεσιών. Πρέπει να βρούμε τρόπου να την επεκτείνουμε, ναι. Είχαμε μια συζήτηση για το μήνα των αφιερωμένων στην ενιαία αγορά και βέβαια οι υπηρεσίε είναι πολύ σημαντικό τμήμα τη όλη διαδικασία. Πρέπει κάπω να το προωθήσουμε μάλιστα ίσω. Κυρία Κοράτσα Μπίλ, μήπω θέλετε να συνοψίσετε και να μα πείτε το χρονοδιάγραμμά σα. Κύριε Πρόεδρε, να αρχίσω από αυτό που είπατε. Γιατί είπατε με πάρα πολύ καλό και σαφή τρόπο ποιο είναι το βασικό μήνυμα της έκθεσής μας δεν είναι μόνο νομοθετικό θέμα. Ε, πρέπει να είναι ένα πολιτικό θέμα, να είναι, να είναι καταλήτης της οικονομίας ε, η εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Ξέρω ότι θα είστε πολύ καλός πρέσβης μας, ε, όπως πάντοτε είστε, για το πρόγραμμα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Θα ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία, να τα διευκρινίσω μάλλον, σε σχέση με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κυρία Γκέπχαρτ. Χαίρομαι που υπάρχει τόσο πολύ σύγκληση για τα θέματα, για το στόχο και την ουσία της έκθεσης αυτής και το θέμα της διάκρισης κατά των καταναλωτών, ότι είναι κάτι το απαράδεκτο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στο άρθρο 20 εδάφιο 2 δεν θέλω να υπονοήσω ότι υπάρχει υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να πολλούν το λέω στην αιτιολογική μου έκθεση, ίσως θα το καταστήσω σαφέστερο μέσω τροπολογίας, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Χαίρομαι που είπατε ότι είναι περιορισμένη η έκθεση σε σχέση με το πόσους χαρακτήρες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, οπότε θα ήθελα όλους να σας ζητήσω να επικεντρωθείτε στην ουσία της έκθεσης, γιατί δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Και χαίρομαι κυρία Γκέπχαρτ που αναφερθήκατε στη σχέση ανάμεσα στο άρθρο 20 και στο άρθρο 1 που λέει ότι το εργατικό δίκαιο είναι ένα εθνικό ε, θέμα και δεν είναι τμήμα του πεδίου εφαρμογή τη έκθεσης αυτής. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο θέμα του συναδέλφου από τους φιλελευθέρους. Α, μήπως το κάλυψα. Ναι, ούτως ή άλλως για το άρθρο 20 μιλήσατε κι εσείς, το κάλυψα άρα. Όσον αφορά τώρα αυτό που είπατε για την εθνική νομοθεσία, να σας πω το εξή. Εγώ δεν λέω ότι η εθνική νομοθεσία είναι λάθος, ούτε είπα ότι δεν θέλω να έχουμε εθνική νομοθεσία, για όνομα του Θεού. Είπα απλώς ότι θα ήθελα να εφαρμοστεί μία οδηγία υπηρεσιών με τρόπο που να είναι ε, συνεκτικός ε, ε, και να εντάσσεται στην εθνική νομοθεσία. Τουλάχιστον να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση. Αυτό τουλάχιστον μπορούμε να το πετύχουμε και νομίζω ότι τουλάχιστον γι' αυτό συμφωνούμε. Για την κυρία Ρούλε θα ήθελα να πω, έχουμε πολύ χρόνο. Μην ανησυχείτε. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 7 Μαΐου. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στις 29-30 Μαΐου, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ε, τον Ιούλιο και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβρη. Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να, να τιμωρήσουμε τα κράτη-μέλη. Ναι, βεβαίω, αυτό συμφωνώ. Εμένα η έκθεσή μου είναι πρόσκληση σε διάλογο. Δεν θέλω να τιμωρήσω κανέναν. Ναι, να δουλέψουμε μαζί με συστάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αναθεώρηση ομοτήμων, ε, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε όλα τα δυνατά φόρα. Μαζί και με την Ιρλανδική Προεδρία βεβαίω, για να δούμε πού μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει με κατευθυντήριε γραμμέ για να εφαρμοστεί η νομοθεσία αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, δεν θα έπρεπε λόγοι δημοσίου συμφέροντος να χρησιμοποιούνται για να μην εφαρμόζεται η νομοθεσία και για να μην δίδεται αυτή η νέα όθηση που χρειάζεται λόγω της κρίσης και λόγω του ιστορικού ποσοστού ανεργίας που έχουμε τώρα στην Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε, νομίζω, επικοδομητικά το ζήτημα αυτό. Ε, αποκινούμε τα κράτη-μέλη Ελπίζω να απάντησα σε όλα τα σχόλια. Αν όχι, παρακαλώ να μου το πείτε. Να σας ευχαριστήσω όλους, τον Διερή, ε, τη Γραμματεία, ε, τους κοιόδης εισηγητές και εσάς τον ίδιο κύριε Πρόεδρε για την υποστήριξή σας. Θα φύγω από εδώ πιστεύοντας ότι είμαστε όλοι, ε, έχουμε όλοι την ίδια άποψη. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσουμε πρόοδο μέσω τη εκθεσή τη. Είναι σημαντικό να έχουμε μια θέση του Κοινοβουλίου πριν από την ε, διάσκεψη, από την Σύνοδο ε, Κορυφής για την Ανάπτυξη, το φθινόπωρο. Το συζητούμε κάποιο, το συζητάμε ήδη πολύ καιρό. 7 Μαΐου λοιπόν για τις τροπολογίες, 29-30 Μαΐου εξέταση αυτών. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τον Ιούλιο και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβρη. Έτσι προτείνω. Ναι. Συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τελευταίο το θέμα αυτό για σήμερα είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή ε, Βιομηχανίας η κυρία Φερχάιν δυστυχώ όμως ε, αποσιάζει, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Ε, θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Ξέρω ότι υπάρχει ένα θέμα συμβαστικών γιατί είμαι σκιώδης. Ο κύριος Μπίνεκολς είναι εδώ και ο κύριος Λέκεργαρτ έφυγε. Α, ξέρω κάπου εδώ είναι, τον είδα πριν. Ο κύριος Έγκστρομ αποσιάζει. Από την Επιτροπή ποιος είναι εδώ. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είδα. Α, θα ακούσουμε αργότερα όταν θα προσέλθει ο αρμόδιος υπαλλήλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τώρα. Ο Ζουβέ να μας τα πει που εκπροσωπεί την εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εισηγήτρια δεν ήταν δυστυχώς διαθέσιμη για να συμμετέχει σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για το σύννεφο και... Ε, για, και γι' αυτό είδαμε πολλές τροπολογίες έχουν κατατεθεί, ε, πολλές ε, σημαντικές, ε, σημαντικά θέματα όπως η προστασία των στοιχείων, η προστασία των καταναλωτή σε σχέση με το σύννεφο και τα περισσότερες τροπολογίες έχουν κατατεθεί από την ίδια την εισηγήτρια. Μετά από μια πρώτη συνάντηση των σκιωδών στο Στρασβούργο έχουμε καταρχήν την μεγάλη ταχύτητα. Η κυρία ε, Φερχέιν θεωρεί πως είναι απαραίτητο αυτό για την ανάπτυξη του σύννεφου. Ε, ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ίντερνετ για όλους τους πολίτες. Δεύτερον, η δυνατότητα ε, πρόσβασης ε, και δυνατότητας μεταφορές, ε, η, υπολογιστικού νέφους να μην περιορίζουν τους καταναλωτές, τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών και να μπορούν να τα μεταφέρουν μέσα σε μια λογική προθεσμία. Αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία του καταναλωτή. Σαφείς απαιτήσει για την ύπαρξη μεταξύ απαιτήσεων και συμβατικών όρων, ώστε να αποφευχθούν οι καταχρηστικές πρακτικές να ενημερώνονται δε οι καταναλωτές για τις υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους πλήρως και ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ένωση. Τέταρτο σημείο αφορά τις, το, το, το, τους όρους, τους συμβατικούς όρους, τους χαρακτηριστικούς. Χαιρετίζονται οι πρόοδοι της Κομισιόν ώστε να υπάρχουν όροι, τι, μάλλον ε, τυποποιημένοι όροι σε ολόκληρη την Ένωση, πράγμα που δεν πρέπει να εμποδίσει όμως την αγορά να συνεχίσει να αναπτύσσει τις υπηρεσίες ε, του σύννεφου. Η, τέλος, υποστηρίζεται τις τροπολογίες του κυρίου Χάρμπορ που στηρίζουν τη δημιουργία μιας προσέγγισης τεχνολογικά ουδέτερης, διαλειτουργικής και ανοιχτής, έτσι και πάλι να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και η προστασία του καταναλωτή. Επόμενο σημείο, η προστασία των δεδομένων και μεταφορά των δεδομένων σε τρίτη χώρα στηρίζει την προσέγγιση που εγώ ο ίδιος Ανέπτυξα σε τροπολογία που κατέθεσα την υπαριθμό 51, όπου δηλαδή μπορεί να υπάρξει πρόβλημα καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς και τον καθορισμό, του καθορισμού της ευθύνης κάθε μέρους, γιατί υπάρχουν εταιρείε που αποθηκεύουν τα δεδομένα σε τρίτες χώρες και η σχετική νομοθεσία θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε κάθε μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς μια τρίτη χώρα να γίνεται μέσα στο σεβασμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ε, χρήση των δεδομένων και την προστασία αυτών. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνεται ο καταναλωτής από τη στιγμή που η εταιρεία που χρησιμοποιεί κοινοποιεί τα στοιχεία αυτά ή τα αποθηκεύει σε τρίτη χώρα. Έπειτα, θεωρούμε πως η Κομισιόν πρέπει να, να αποφασίσει και για την δυνατότητα προώθησης της δημιουργικότητας προς όφελος των δικαιούχων, πνευματικών δικαιωμάτων και των χρηστών. Τελευταίο σημείο είναι ε, το τέλος για ιδιωτική ε, αντιγραφή. Ε, θα πρέπει και αυτό να αναφέρεται μετά από τη δημοσίευση της έκθεσης του κυρίου Βιτορίνο. Ε, θα πρέπει δεν να συνάπτονται συμφωνίες αδειοδότησης ε, αλλά χωρίς να επιβάλλονται νέα τέλη μέσω της ε, εφαρμογής για το υπολογιστικό νέφος ή την χρήση αυτού. Αυτά είπαν οι και ελπίζω πως μεγάλη πλειοψηφία θα συστηρίξει τις συμβαστικές. Ε, αν μπορώ να έχω το λόγο για λίγο... Ευχαρίστω για να εκφράσω τη δική μου άποψη, εκτός και αν μπορώ να το κάνω τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Θέλω να παραθέσω την 22 για την έννοια της δυνατότητας μεταφοράς των στοιχείων, το είδος των στοιχείων δηλαδή που πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν ε, πολύ ομαλά αν κανείς αλλάξει ε, πάροχο. Έπειτα Το υπολογιστικό νέος πρέπει να θεωρηθεί ω μια δυνατότητα για ανάπτυξη, ανάκαμψη τη ευρωπαϊκή οικονομία και έπειτα ήθελα να μιλήσω για την στρατηγική θέση τη πραγματική τοποθεσία των κέντρων αποθήκευση ή συλλογή των στοιχείων και τη δυνατότητα εγώ ας πούμε ως, ως ε, δεν θα ήθελα τα στοιχεία μου να αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων που ε, στην ουσία βρίσκονται στην Κορέα ή στην, στην Νότια Κορέα ή στην Κίνα. Αν ήμουν στρατητικός, ας πούμε δεν θα ήθελα τα δικαιώματα, τα στοιχεία μου να αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων που ε, βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα. Π.χ. δύο-τρία παραδείγματα που σας δείχνουν εύγλωτα την σημασία του, του πραγματικού τόπου αποθήκευση αυτών των δεδομένων. Thank you very much. Uh, ευχαριστώ, κύριε Βάιντενχολτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια πάρα πολύ. προσπάθησε να ανταποκριθεί σε όλες τις ε, τροπολογίες και πάντα ε, με συνενετικό πνεύμα τα συζητούσε μαζί μας. Η δυνατότητα μεταφοράς των ε, στοιχείων για των δεδομένων είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και οι εγγύησεις για την προστασία των δεδομένων επίσης. Και να μην παρουσιάζεται αυτό σε εμπόδιο ή βάρος αλλά στο cloud ε, είναι και συγκριτικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικό για την Ευρώπη. Θα μπορούσαν κάποιοι να φέρουν τα δεδομένα τους στο ευρωπαϊκό νέφος. Επίσης, η ουδετερότητα του δικτύου είναι πάρα πολύ σημαντική, με ελευθερία πρόσβασης εννοώ. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση αυτή και μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση προς μια περαιτέρω ενοποίηση της στρατηγικής μας στην Ευρώπη για το cloud computing, το υπολογιστικό νέφος. Ο κύριος Λέκεγκαρτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αφού απουσιάζει η συγγήτρια θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ σύντομος. Ευχαριστώ πολύ. Διάβασα τις τροπολογίες με μεγάλο φυσικά ενδιαφέρον. Ε, το υπολογιστικό νεφό ναι, στο μέλλον θα είναι από τους φορείς ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, δεν χωρά καμία αμφιβολία. Και αυτό ε, που παίζει ρόλο είναι το να έχει κανείς δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ε, θα ήθελα και πάλι να εκφράσω τη λύπη μου για τα κράτη-μέλη που ζήτησαν να περικοπεί η διευκόλυνση Connecting Europe, διασυνδέοντας την Ευρώπη. 8,2 δισεκατομμύρια έκοψαν. Μα πώς θα διασυνδέσουμε την Ευρώπη και πώς θα συνδεθούμε όλοι στο διαδίκτυο με τέτοιες περίκοπες. Και πώς θα έχει στο μέλλον υπολογιστικό νέφος αν δεν υπάρχει καν σύνδεση στο διαδίκτυο. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η συγγήτρια. Χαίρομαι που βλέπω να υπάρχει γενικότερη συνένεση στα βασικά θέματα μεταξύ των πολιτικών ομάδων και θα κάνουμε και συμβασμού. Προσβλέπω λοιπόν στην καλή συνεργασία με την συγγήτρια και σα ευχαριστώ. Ε, η κυρία Ρούλα. Και εγώ πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πραγματικά έχει συνοψίσει τα σημαντικότερα στην έκθεσή της, αλλά και με δικές της τροπολογίες έχει κάνει κάποιες συμπληρώσεις. Οπότε για μας είναι περιττό να κάνουμε οποιασδήποτε τροπολογίες για την προστασία των δεδομένων. Ε, τα έχει χειριστεί όλα αυτά πάρα πολύ καλά, ικανοποιητικά και η έκθεση θα είναι καλή. αυτή η Επιτροπή, η δική μας δηλαδή, είναι αρμόδια και για τα δικαιώματα των καταναλωτών και αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονούμε ούτε σε αυτό το θέμα. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και εγώ ήμουνα εισηγητής ε, του Κοινοβουλίου για την Καθολική Υπηρεσία τα Δικαιώματα των Καταναλωτών στην Οδηγία για τις Τηλεπικοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αντίστοιχα θα ισχύσουν εδώ και στο cloud computing. Αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε πώς οι καταναλωτές πλέον χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες υπολογιστικού τους νέφους ε, και με, έναν τρόπο που είναι φαινομενικά ε, απρόσκοπτος. Τώρα δεν ξέρω αν έχει δίκιο ο κύριος Ζουβένα, θα πρέπει να θορυβήσουμε τους ε, καταναλωτές και να αρχίσουν να ανησυχούν για το πού φυλάσσονται τα δεδομένα τους. Αυτά είναι θέματα διεθνή, έχουν να κάνουν με την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια. Θα αρχίσουμε να το συζητάμε αυτά σήμερα το απόγευμα και θα πρέπει να το δούμε σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικές επίσης και επικείμενες εμπορικές συζητήσεις που θα γίνουν διεθνώς. Πρόσφατα πήγα να αγοράσω μία κάμερα και πολλές, ε, και μία φωτογραφική μηχανή μάλλον, ε, συνδέονται άμεσα με το διαδίκτυο. Δηλαδή, μόλις βγάζεις μια φωτογραφία, βγαίνει αμέσως στο ασύρματο ε, και πάει στο cloud σου, στο συνεφάκι σου. Και με ρώτησαν όταν αγόρασα τη φωτογραφική μηχανή αν θέλω να αγοράσω αμέσω και το υπολογιστικό νεφο. ταυτόχρονα. Είναι η άμεση προσφορά. Ναι, αλλά ποιε είναι οι προποθέσει και ποιοι είναι οι όροι που ισχύουν. Και πώ γίνεται αυτό τόσο αυτόματα, διακτηνίζεται η φωτογραφία από τη φωτογραφική μηχανή και πάει κατευθείαν στο νέφος με την κινητή ε, τηλεφωνία το θέμα τη φορητότητα του τηλεφωνικού αριθμού. Θυμάστε το συζητούσαμε ε, στις τηλεπικοινωνίες πολύ αυτό. Λοιπόν, τι ισχύει αυτό, ποιε είναι οι υποχρεώσεις, οι όροι που ισχύουν, τι υπογράφεις όταν δέχεσαι ένα τέτοιο νέφος και ποιε είναι και οι συμβατικές σου υποχρεώσεις. και πώς θα μεταφέρονται τα δεδομένα, ας πούμε, θες να αλλάξεις πάροχο, προμηθευτή, ε, για να αποθηκεύονται σε άλλη εταιρεία. Αυτό πώς θα γίνει. Ε, χρειάζονται διάφορες εγγύησεις και ε, προϋποθέσεις να προσεχθούν. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη πραγματικά και εύστοχη αυτή η πρόταση και καλό είναι εμείς να τη βελτιώσουμε. Ένα άλλο σημείο την περασμένη εβδομάδα συνεργάστηκα με τον κύριο Έγκστρομ για συμβαστικές τροπολογίες και αξίζει να το πούμε. Μπορεί να μην είναι η άμεση αρμοδιότητά μας, αλλά επασχολεί πολύ τους καταναλωτές αυτό το θέμα του copyright, τα πνευματικά δικαιώματα. Και τι ε, διαπνέει από τις, διαπνέει τις ε, τροπολογίες του κυρίου Έγχομ. Είτε πρόκειται για μουσική, είτε πρόκειται για βίντεο. Μπορεί κανείς να θέλει ε, να το χρησιμοποιήσει ή να το αποθηκεύσει απλώς στο υπολογιστικό του νέφος. Και τι θα γίνει με τα τέλη, ας πούμε. Δεν μπορεί να χρεώνεις επιπλέον ακριβώς επειδή κάποιος ακούει ένα προϊόν και με ένα διαφορετικό τρόπο θέλει να το μοιράζεται θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ο κύριος Μπαρνιέ το εξετάζει αυτό το καιρό στις υπηρεσίες του, εκπονούν αντίστοιχα έγγραφα, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη εστίαση σε αυτό το θέμα. Επιταχύνονται οι εξελίξεις, γιατί επιταχύνονται και οι δυνατότητες πρόσβασης και πώς χρησιμοποιεί ο κόσμος ε, τις συσκευές ε, και τα διάφορα που υπάρχουν πλέον ως δυνατότητες αποθήκευσης δεδομένων. Πολύ σύντομα θα καταθέσω συμβαστικές τροπολογίες και περί τα τέλη Μαΐου προβλέπω να γίνει η ψηφοφορία. Ποιος θέλει το λόγο. Α, η κυρία Γκαλό για το copyright, για τα πνευματικά δικαιώματα. Όχι, όχι, δεν θα μιλήσω εγώ για το copyright. Ε, γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε ότι τα θέματα αυτά τα ψηφιακά με συναρπάζουν και μου εξήγησαν πάρα πολύ λεπτομερώς TST Cloud Computing. Και πρέπει να σας πω ότι ε, ε, ο χώρος όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα, σε αντίθεση με τα όσα είπε ο ξέρετο συνάδελφος Φιλίπ Ζουβά, ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα δεν είναι καθόλου καθοριστικός η τοποθεσία. Αυτό που έχει σημασία είναι το λογισμικό πρόσβασης ή ανάκτησης αυτών των δεδομένων, ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Ε, που δεν έχει σημασία και ο έλεγχος που θα πρέπει να κάνουμε δεν είναι που βρίσκονται σε ποια χώρα ή σε ποιο σημείο, είναι πώς θα τα ανακτήσουμε και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα ή πώς θα τα δώσουμε σε άλλον πάροχο ή σε άλλον προμηθευτή, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει μια σύγχυση εδώ. Δεν έχει σημασία, ας πούμε. Ε, και όταν γίνεται λόγος για κυρίαρχο cloud, εθνικό cloud. Τι σημαίνει αυτό, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη είναι κέντρα επεξεργασία για να έχουμε τον έλεγχο των δεδομένων. Τώρα αν αποθηκεύονται γεωγραφικά στην Κίνα δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μπορούμε να τα φέρουμε εδώ, να τα χρησιμοποιούμε όπως ε, φρονούμε. Αυτή ήταν η μόνη μικρή ε, τεχνική εξήγηση που ήθελα να σας δώσω, γιατί ε, αφιέρωσα πολύ χρόνο σε αυτά τα θέματα. Ξαναφεύγω αύριο για τις Ηνωμένε Πολιτείες για να δω τι γίνεται εκεί, εκεί σε πολύ σημαντικές εταιρείες, ε, παρόχους. Ε, τώρα δεν θα πρέπει να έχουμε φαντασιώσεις ε, και να ζούμε σε ένα φανταστικό κόσμο έτσι με τα συννεφάκια, να δούμε πώς είναι η τεχνική πλευρά του θέματος και μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Καπαλάγκο είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να της δώσω το λόγο. ο κύριος εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μας δίνετε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια ε, σύντομα σχόλια. Διαβάζοντας τις τροπολογίες θα λέγα ότι είναι πάρα πολύ θετική ε, η εντύπωση που έχουμε για την ανταπόκριση των μελών της Επιτροπής σας ε, σε σχέση με το υπολογιστικό νέφος. Η προσέγγιση, μας, ε, η προσέγγιση είναι πολύ θετική σε σχέση με το νέφος. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει σε στάδια να γίνει πιο φιλική προς το υπολογιστικό νέφος. Ε, αποτελεί τουλάχιστον ένα ορόσημο αυτό για μας, σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Ε, και ε, συμφωνώ απολύτως με τα περισσότερα, εξ είπε ο Φιλίπ Ζουβά, εκ μέρους της εισηγήτριας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το θέμα της ε, βριζονικής υποδομής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί βεβαίως ε, με τα σχόλια για τη διευκόλυνση που για την ώρα δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες που είχαμε ε, προς, την, προς, προς το, όταν υποβάλαμε το αίτημά μας προς το Συμβούλιο. τα επικουρικά αλλά και τα κύρια δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά, ως προς την πρόσβαση εννοώ σε αυτά, ώστε να έχουμε μία ε, ε, πρόσβαση ε, και μέσω των ε, συστημάτων, των κινητών συστημάτων επίσης. Όσον αφορά τις συμβατικές ρήτρε, το νομικό πλαίσιο, με όλες τις ε, προσπάθειες που γίνονται για την προστασία των δεδομένων και την παρακολούθηση, ό,τι έχει να κάνει με το ιδιωτικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικά για μας και ε, τα επικροτούμε απολύτως. Μου άρεσε ας πούμε το ερώτημα του, της διατήρησης ενός αντιτύπου της μουσικής, για παράδειγμα, σε κάποιο σημείο του, νε, του νεφους, κάτι που ανεφέρατε και εσείς εμέσως, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι. Έχουμε συγκεκριμένη εταιρική σχέση που την ιδρύσαμε για να υπάρξει προϋπολογισμός ώστε να είναι υψηλότερη χρήση του νεφους, ειδικότερα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όσον αφορά τώρα ε, το πού βρίσκονται τα κέντρα δεδομένων, ε, οι πτυχές ε, που αναφέρθηκαν μπορούν να αντιμετωπιστούν και με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δυναμικού στην Ευρώπη και περνά μέσα από ισχυρούς φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα αυτό. Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία των δημοσίων προμηθειών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο ε, στην πλευρά της προσφοράς ε, που θα πρέπει να είναι πιο ε, πλήρης στην Ευρώπη, πιο πλούσια στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε μόνο μεγάλους φορείς, γιατί για την ώρα αυτοί δεν παρέχουν καλή, καλές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Για πιο καινοτόμες λύσεις θέλουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης και την ιδιωτική αγορά όσον αφορά την προσφορά να μην μιλήσω για το περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορεί να επωφεληθεί από τον έφος και τους καταναλωτές βέβαια. Υπάρχει πτυχή των προδιαγραφών, υπάρχει πτυχή ε, ε, του επίπεδου των υπηρεσιών και των πιστοποιήσεων ε, και ούτω καθεξής. Είμαστε λοιπόν σε μια πολύ βαθιά συζήτηση, διεξοδική, εμείς με πολύ χαρά θα εξετάσουμε τις τροπολογίες ε, και θα σας υποστηρίξουμε σε ό,τι, σε ό,τι μπορούμε από πλευράς μας κυρίως για τις πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν όσον αφορά την ε, ε, βελτίωση της ανακοίνωσης. Θα καταλάβετε, επειδή όλη η διαδικασία ξεκίνησε 27 Σεπτεμβρίου του 2012, είμαστε στη μέση μιας μεγάλης διαδικασίας με τον κλάδο, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τις δημόσιες αρχές, τους καταναλωτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε για τη συμφωλή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε τι δυνατότητες μπορούμε να έχουμε ε, για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, μας είπε ο Φιλίπ Ζουβέ ορισμένα πράγματα, ήδη εκπροσωπώντας την εισηγήτρια. Έχουμε ήδη κάνει μία συνάντηση με τους ε, σκι, σκιώδεις εισηγητές και με την κυρία Φερχόιεν. Ελπίζω ότι θα έχουμε συμβαστικές τροπολογίες που θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Θα γίνει τον Οκτώβριο του 2013, αργή ακόμα, Νοέμβριο θα περάσει από την Ολομέλεια. Ίσως θα μπορούσαμε λίγο να τα επιστέψουμε τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας για σήμερα το πρωί. Να σας υπενθυμίσω ε, όσοι δεν ε, βλέπετε, μας βλέπετε στο ίντερνετ και δεν έχετε δει ακόμη το ενημερωτικό μας ε, φυλάδι, δεν έχετε εγγραφή, μπορείτε να το κάνετε. Σήμερα το απόγευμα θα ε, έχουμε τη συζήτησή μας ε, για τον κυβερνοχώρο και τη στρατηγική ασφαλείας. Είμαστε αρμόδια επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σήμερα το... τη μελέτη αντικτύπου για τη στρατηγική αυτή. Τέσσερις η ώρα. Θα σας περιμένω λοιπόν και τους συναδέλφους εδώ αλλά και στο διαδίκτυο, όποιον θέλει να παρακολουθήσει. Πολύ σημαντικές προτάσεις έχουμε και για τα ιατροτεχνικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Θα αρχίσουμε τρεις η ώρα με το θέμα αυτό. Θα λέμε λοιπόν το απόγευμα και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα το πρωί.